Λοιπόν, καλημέρα σας. Μου λένε πως το ρολόι αυτό είναι και 5 λεπτά πίσω. Ίσως να είναι λιγότερο. Δεν είναι εδώ όλοι οι ισχυώδεις εισηγητές για το πρώτο θέμα στην μυρίσια διάταξη. Να κάνω τις ανακοινώσεις της Προέδρου που αναβλήθηκαν από χτες. Λίγα πράγματα από την δεύτερη δόση του τριμερούς διαλόγου. Η πρώτη έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο και κάλυψε τα βασικά ζητήματα που είχαμε δει εκ των προτέρων. Συμφωνήσαμε σε κάποιους συμβασμούς, σε κάποια τεχνικά θέματα, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει. Το Συμβούλιο δεν έχει απαντήσει στο βασικό ε, ζήτημα που είναι η, ε, καταληκτική ημερομηνία. Και βεβαίως αυτές έπρεπε να αναβληθεί ο τριμερής διάλογος καθώς ε, ταυτόχρονα ε, υπήρχε και διάλογος για ένα άλλο θέμα για τον ΕΜΙΡ. Για τις ακάλυπτες ε, πωλήσει, η τελευταία συνάντηση τριμερής έγινε στις 5 Οκτωβρίου και πάλι είχε αφιερωθεί σε συζητήσεις για το άρθρο 12β ασφαλιστά κινδύνου για κρατικά ομόλογα και Ε, υπάρχει κάποια πρόοδος, αναμένουμε μια επιβεβαίωση για το πότε θα είναι όλοι έτοιμοι για την επόμενη συνάντηση, πιθανώς την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν από τις τριμερείς συναντήσεις. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής. Και ο εισηγητής μας είναι ο Ανδρέας Σβάμπ και θα εξετάσουμε τώρα τις ε, τροπολογίες. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν ε, τροπολογίες και επικοδομητικές ε, προτάσεις, ειδικά τους σκιώδεις εισηγητές, σαν Σεσπρεσέδο, Έπινγκ και οι υπόλοιποι δεν έχουν έρθει ακόμα. Ήδη μπορούμε να δούμε από τώρα πως υπάρχει ευρία συμφωνία σε πολλά ζητήματα. Η ευθύνη της Επιτροπής μας είναι κατά την άποψή μου πως ε, θα πρέπει να ε, αναφέρουμε και να συμπληρώσουμε τα ζητήματα τα οποία είναι κέρια για τον ανταγωνισμό, για την Επιτροπή ε, Νομικών Θεμάτων και να γίνεται βεβαίως η επιβολή της ε, νομοθεσίας μέσω της Κομισιόν, μέσω προστήμων. Μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία πρέπει να παραμείνει έτσι. Όταν μιλάμε λοιπόν για συλλογική προσφυγή στην Ευρώπη, θα πρέπει να προσφέρουμε ασφάλεια δικαίου και βεβαίως ε, αποσμιώσεις οι οποίες θα βασίζονται σε μια στιβαρή νομική και τελικά κοινωνική βάση. Πρέπει να διατηρηθεί βέβαια στο δίκαιο του ανταγωνισμού και να μην έχουμε όλες τις αρνητικές συνέπειες που είχε σε άλλες χώρες η λογική προσφυγή. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνω πως ή ε, έχουμε αρκετά σημεία σύγκληση κάτι το οποίο δεν συνέβαινε εξ Αυτό συμβαίνει νομίζω και λόγω των ε, διαφόρων συμβαστικών ε, τροπολογιών. Π.χ. από τον συνάδελφο Σάντσε Πρεσέδο υπάρχουν σε μια τροπολογία, μια σειρά δικλείδες ασφαλείας, ε, τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πριν καταλήξουμε στην νομοθεσία και νομίζω πως ταιριάζουν πάρα πολύ με αυτά τα οποία είχα πει και εγώ λίγο πολύ και άρα συμφωνούμε. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω πως πρέπει επίσης να είναι σαφές πως για τη ρύθμιση αυτών των δικλειδών δεν μπορούμε και δεν έχουμε στο Κοινοβούλιο όλες τις ε, νομοθετικές αρμοδιότητες άρα θα πρέπει να γίνει αυτό στο επίπεδο των κρατών μελών. Η συμβαστική γραμμή λοιπόν στο πρώτο θέμα που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει με το οριζόντιο οριζόντια αριθμισή για να παρουσιαστεί στην ε, κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή πριν τα Χριστούγεννα. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οπωσδήποτε μορφή της ε, συλλογικής προσφυγής αλλά και να πούμε πως ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν προσφέρεται παρά μόνο σε περιορισμένο βαθμό για μια ενιαία προσέγγιση γιατί βεβαίως υπάρχει ήδη μια ε, δημόσια διαδικασία επιβολής την οποία δεν θα πρέπει να εξασθενήσουμε αλλά να την ενισχύσουμε πρώτον αυτό και δεύτερον γιατί θα πρέπει να δούμε και τις ιδιαιτερότητες οι οποίες υπάρχουν ήδη στο δίκαιο του ανταγωνισμού και θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μια μέση οδός, αλλά νομίζω πως θα καταφέρουμε σε αυτή την γνωμοδότηση. Και προτείνω εγώ εδώ πέρα και περνάμε στο δεύτερο θέμα να δούμε ποιες θα τι θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δώσουμε τη συνέχεια στον κάθε κλάδο χωριστά γιατί εδώ πέρα είναι σαφές πως ε, η Κομισιόν ε, όσον αφορά την ε, δημόσια δικασία. Έχει ολοκληρώσει την ε, εργασία της, καθώς επίσης και όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Κομισιόν. Και με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια. Όμως αυτό είναι κάτι το διαφορετικό από τις ε, λεγόμενες ε, ιδιωτικές κινήσεις που να γίνουν όπως λέμε και στις υπόλοιπες ε, περιπτώσεις γιατί όπως σας είπα βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο μιας δημόσιας διαδικασίας και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στις περιπτώσεις παραδείγματο χάρη όπου, στις περιπτώσεις όπου οι ενάγοντες έχουν μια απέτηση για δημοσιοποίηση κάποιων ε, εγγράφων. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τις δύο περιπτώσεις και να πούμε πως η λεγόμενη private action είναι κάτι το οποίο μπορεί βεβαίω να απασχολήσει την ε, Κομισιόν, αλλά δεν αφορά ιδιαίτερα την Επιτροπή μας, αλλά οτιδήποτε βεβαίω ε, αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού οπωσδήποτε. Τώρα για τις μπικλίδες ε, ασφαλείας, δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Τέλος για το τέταρτο αυτό σημείο του συμβασμού για τις εναλλακτικέ μορφές επίλυσης διαφορών θα πρέπει να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε κάποιον να καταφύγει σε αυτές εάν δεν το θέλει. Νομίζω λοιπόν πως ε, σας ανέφερα τα σημεία τα οποία ακόμα εκκρεμούν και το θέμα λοιπόν είναι ακόμα ανοιχτό το τι θα κάνουμε με τις ε, private actions, εάν θα τις ενσωματώσουμε εδώ πέρα ή εάν θα μείνουν χωριστά σε ένα οριζόντιο μέσο. Αναμένω λοιπόν να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι και σας ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τη γραμματεία, κυρία Πρόεδρε. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τους δεν λύνουν πρώτα. Muchas eh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τον κύριο Σβάμπ, απαντώντας... στο ίδιο πνεύμα διαλόγου για την επιτυχία συμφωνίας όσον αφορά τις συλλογικές ε, αυτές εκκυρώσεις, επεξήγησε τέλεια ποια είναι τα θέματα υποσυζήτηση. Πρώτο, το αν πρέπει να υπάρχει ή όχι ένα οριζόντιο ε, μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση που πάντα είχαμε είναι ότι χρειαζόμαστε μια ε, οριζόντια εστίαση. Αυτή η οριζόντια εστίαση για την αντιμετώπιση όλων των συλλογικών αυτών θεμάτων θα επιτρέπει να υπάρχει ένα σύλλογο θεμάτων στον τομεακό τομέα που θα εφαρμόζονται, αλλά υπό το πρίσμα του δικαίου για τον ανταγωνισμό, εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία προέρχεται και έχει νομικές βάσεις. Η νομική βάση για τον ανταγωνισμό είναι μια διαφοροποιημένη νομική βάση. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία προηγούμενη που θα εφαρμόζεται σε σχέση με το δίκαιο για τον ανταγωνισμό. Και έτσι η Επιτροπή Οικονομίας ή οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις ουσιώδεις ε, πτυχές ε, του ανταγωνισμού θα έπρεπε να ασχολούνται με αυτές. Συμφωνούμε να υπάρχει οριζόντια εστίαση, αλλά πρέπει να δούμε και τις ιδιομορφίες και τις, ε, την ιδιοσυστασία του δίκαιου για τον ανταγωνισμό. Έχουμε εδώ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, η πολιτική για τον ανταγωνισμό και το δίκαιο για τον ανταγωνισμό πάντα έχουν σε σχέση με τη συνθήκη την αποτελεσματικότητα ως στόχο της πολιτικής του ανταγωνισμού. Το εγχείρημα δηλαδή, η, άσκηση εξουσιών από τις αρχές ε, αρμόδιες ε, για τον ανταγωνισμό είναι σημαντική υπόθεση. Πρέπει να αρθρώνεται λοιπόν μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αυτό το θέμα και να υπάρχουν κριτήρια ώστε ο δημόσιος τομέας να μην αποδυναμώνεται λόγω του ιδιωτικού. Πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο μέτρων και να το δούμε σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Παράδειγμα, προστασία προγραμμάτων, ε, ε, αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις έρευνες, ε, και πώς θα υπάρχει αποτελεσματικό πλαίσιο κυρώσεων. Μέσα στον ανταγωνισμό υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο σε σχέση με εκείνο που υπάρχει σε, άλλα, σε άλλους τομείς του κοινοτικού τομέα, όπως παράδειγμα στην προστασία των καταναλωτών, διότι ο ανταγωνισμός αφορά και τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και αφορά και τις σχέσεις με τους καταναλωτές. Είναι ένα υψηλότερο, σημαντικότερο επίπεδο. Γι' αυτό έχει ιδιομορφίες ο ανταγωνισμός που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Το τρίτο θέμα είναι αν πρέπει να υπάρχουν δράσεις παρακολούθησης ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΔΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των θυμάτων να υπάρξει αυτή η δράση και έτσι λοιπόν από πλευρά ε, του δημόσιου τομέα πρέπει να λαμβάνετε αυτό υπόψη. Ένα άλλο τομέα ε, σε σχέση με το δημόσιο είναι θέματα τα οποία πρέπει ακόμα να επιληθούν. Υπάρχουν δύο δυνατότητε. Δράσει ε, συνέχεια ή παρακολούθηση και αυτόνομε δράσει. Θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα διάρθρωση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Επόμενο ερώτημα. Ποιο θέμα θα υπάρχει το opting in ή το opting out Συμφωνούμε όλοι ότι είναι μια καλή αρχή να αρθούν οι διαφορές σε σχέση με την ε, ε, βόρειο-αμερικανική ρύθμιση, σε σχέση με προσφυγές σε δικαστήρια. Εμείς ε, θέλουμε competition και όχι litigation, όχι δηλαδή προσφυγή 200 δικαστήρια. Για το opting in δεν, υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφοροποίηση είτε θα είναι οι αρχές ε, το Υπουργείο Οικονομικών, είτε εκπρόσωποι των καταναλωτών, πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός. Όμως, σε σχέση με τις ε, ομάδες ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση αυτή, σε σχέση με την εκπροσώπηση των θυμάτων που προσφεύγουν στα δικαστήρια όσον αφορά πρακτικές που ισχύουν σήμερα. Γι' αυτό αυτό το θέμα πιστεύω ότι επίσης μπορούμε να το επιλύσουμε χωρίς ιδιαίτερα περίπλοκα προβλήματα. Και έχουμε θέσει δύο ρήτρε διασφάλισης. Η πρώτη αναγνωρίζεται ήδη από το 10, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίζεται στα θύματα η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και τα ισοδύναμα που ισχύουν στις χώρες τους όσον αφορά το εθνικό δίκαιο. Δεν πρέπει να είναι σε χαμηλότερο επίπεδο το ευρωπαϊκό δίκαιο όσον αφορά τις εθνικές ρυθμίσεις. Η ρήτρα λοιπόν αντιστοιχίας ή αντιστάθμισης είναι κάτι το οποίο έχει να γνωρίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεύτερο, όταν υπάρχει κάποια αναγνώριση, θέσπιση στη, ε, κριτηρίων, δεν μπορεί να είναι στενό κορσέ αυτά τα κριτήρια όσον αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με, την, ε, με τις αρχές αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η δικαιακή αρχή και θα είμαστε ελαστικοί και ευέλικτοι, αλλά σίγουρα με κάθε σαφήνεια και κάθετα θα πούμε ότι το δίκαιο για τον ανταγωνισμό έχει ξεχωριστό πεδίο εφαρμογής, αυτοτελές αυτούσιο πεδίο εφαρμογής και πρέπει να το διασφαλίσουμε και δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ε, περιορισμοί Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπέρ ενός οριζόντιου μέσου, αλλά όχι υπέρ προηγούμενης ρύθμισης που θα καθορίζει ποιες είναι οι διατάξεις για την εφαρμογή αυτών. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Επόμενη Σοφία Σελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαιρετίζω τις παρατηρήσεις του εισηγητή. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τεχνική συμφίση αυτό που συζητάμε, αλλά είναι θεμελιώδης κίνηση ώστε να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά. Προκειμένου να υπάρξει εσωτερική αγορά και εφόσον έχουμε εσωτερική αγορά, θα πρέπει να υπάρχουν και κατοχυρωμένα δικαιώματα του καταναλωτή. Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο, θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν ήδη μέσα για τη συλλογική προσφυγή. Μην ξεχνάμε ότι ο καταναλωτή έχει πάντα δικαίωμα να προσφύγει και ατομικά στο δικαστήριο. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από το μηδέν. Κάτι πάνω στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν όλοι είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, όλη διαδικασία. Είτε είμαστε υπέρ μιας μετριοπαθούς έναρξης ή ε, της θέσπισης ενός ευρύτερου μέσου. Φαίνεται όμως ότι γενικά υπάρχει συνένεση σε όλες τις πολιτικές ομάδες και αυτό είναι πολύ θετικό. Νομίζω ότι επίσης φαίνεται να συμφωνούμε πάνω στην ανάγκη για διασφάλιση και για την αποφυγή υπερβολικών δικαστικών διενέξεων, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, όπως έχουμε δει στη ΣΥΠΑ. Με μεγάλη χαρά επίσης άκουσα τις παρατηρήσεις του εισηγητή πάνω στους εναλλακτικούς τρόπους ε, ε επίλυσης ε, ζητημάτων, γιατί είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν νομικά δυνατόν. Αν αναπτύξουμε όμως καλά, καλά εργαλείο διαιτησία, αν θέλετε, θα μπορεί να αποσυμφορεί το δικαστήριο, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση όμως. Και τέλος πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια παρα... ε, και κάποια εργαλεία παρακολούθησης Συμφωνώ με τον ε, κ. Σάντσες Πρεσέντο ότι βέβαια σίγουρα χρειαζόμαστε πολύ ε, ισχυρά μέσα για την ε, δημόσια εφαρμογή και επιβολή, αλλά δεν μπορούμε βέβαια να αποτρέψουμε την προσφυγή ανθρώπων στο δικαστήριο. Και βέβαια είναι και θέμα αποκάλυψη εγγράφων. Δεν είμαι νομικό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα για να μπορεί κάποιο να προσφύγει. και αρκεί βέβαια οι πληροφορίε οι οποίες δημοσιεύονται να μην είναι ει βάρο είτε δημόσιων υποθέσεων είτε ε, δικαιωμάτων εταιριών, αλλά πάντως ο καταναλωτή πρέπει να έχει πάντα δικαίωμα προσφυγής, προς, συγγνώμη, προσπέλαση στα έγγραφα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι το νομοθέτημα αυτό είναι θετικό για την ολοκλήρωση εταιρική αγορά. Δεν είναι μόνο υπέρ των καταναλωτών και των εταιριών, αλλά για να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο διευκολύνεται και ε, ρέι στην εσωτερική αγορά, στην ενιαία εσωτερική αγορά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, The Camping. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σουάμπ για αυτό το σχέδιο νόμης. Έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες στην αρχική έκθεση ε, της Επιτροπής Νομικών Ζητημάτων, την έκθεση ΛΙΝΕ. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στην έκθεση αυτή. Καταρχά νομίζω ότι θα πρέπει να τεκμηριώσουμε σε ποιο βαθμό ένα, ε, απατείται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο συλλογική προσφυγή σε σχέση με την εξασφάλιση των αρχών αλληλεγγύη, επικουρικότητα. Ακούω και την έννοια τη ε, συλλογικότητα, αλληλεγγύη, συγγνώμη, και την ε, μπερδεύω, αν θέλετε. Επικουρικότητα, εν πάση και αναλογικότητα. Η δημόσια εφαρμογή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ακολουθεί επίση και του κανόνε του εθνικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη. Κατά δεύτερο, το σχέδιο της έκθεσης περιορίζεται σε εκθέσεις όπου υπάρχει παραβίαση ε, δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Όμω ε, ε, κοινοτικό δίκαιο ε, δίνει δυνατότητα προσφυγής οποτεδήποτε ε, παραβιάζεται ο νόμος περί ανταγωνισμού. Και φαίνεται αυτά τα δύο να μην συνάδουν. Η εστίαση πάνω στα, ατομικά δικαιώματα για αποζημίωση κάτω από 2.000 ευρώ είναι λανθασμένη. Πρέπει να είναι και ευρύτερη στάξη, ιδιαίτερα όταν υποφέρουν επιχειρήσει. Άρα η, δεν, με αυτόν τον περιορισμό δεν είναι συμβατή το συγκεκριμένο άρθρο για την μη βλάβη εταιριών. Το δεύτερο που κύριε Σβάμπ είναι ότι περιορίζεται η συνολική δημόσια επιβολή απόφαση σε πλαίσια συλλογική προσφυγή όταν υπάρχει γενική παραβίαση. Γιατί να εισάγουμε τέτοιο περιορισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ή άλλω ε, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να πραγματευτεί όλε τι περιπτώσει. Πρέπει να είναι επιλεκτική. Και τι γίνεται με τους καταναλωτές σε αυτή την περίπτωση, πού βρίσκονται. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ της ε, εξουσίας των παραγωγών και των καταναλωτών. Και πέμπτον, ω ένα αλλακτικό μέσο ε, διένεξ, επίληξη διενέξεων, η συλλογική ε, προσφυγή επίση μπορεί να είναι ε, σε αντιδιαστολή σε σχέση με τους μηχανισμούς, του εθελοντικού μηχανισμού επίλυσης. Ο μηχανισμός θα πρέπει να μένει όμως εναλλακτική συλλογική προσφυγή και να μην είναι προϋπόθεση και τέλος, κυρία Πρόεδρε, προβληματίζω από την όλη διαδικασία. Γιατί η Κίσλεϊν φαίνεται να είναι κάποιο είδου Γερμανό ηγητή επίτροπο, σκιώδη επίτροπο ε, προτού κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίσει να παρουσιάζει την πρότασή της. Αυτή είναι μια μέθοδος της κοινοτική ε, μεθόδου που εγκομιάζεται εδώ ή είναι μια ε, επίδειξη, αν θέλετε, κάποιας ε, ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να κάνει σχετική έρευνα και να δώσει σχετικέ εκθέσει και όχι προκαταρτικά να εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα που φαίνεται ο κ. Λίνιν είναι εξοικειωμένο με αυτά, ενώ φαίνεται να αγνοεί τα δικαιώματα εκατομμυρίων καταναλωτών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω. Δεν ε, μπορώ να σα απαντήσω όσον αφορά τη διαδικασία. Ε, είμαι σίγουρη πως η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, ναι. θα σκέφτηκε πως θα ήθελε να ξαναυποβάλει την άποψη. Δεν βλέπω κανέναν από τους πράσινους εδώ πέρα. Γιούργεν, θέλετε τον λόγο για την ΚΟΕ. Όχι κανένα σχόλιο σήμερα. Εξάλλου περιμένει και ο κύριος Τρισέ ήδη. Ε, σας ευχαριστούμε. Ανδρέας. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις επικοδομητικές ε, συνεισφορές ε, των συναδέλφων. Σύντομα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Έπινγκ. Η πρότασή μου για να δοθεί κάποια συνεχεία δεν προβλέπει πως θα καταργηθούν οι ε, ιδιωτικές ε, προσφυγές. Απλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μία μετριοπαθή προσέγγιση στον τομέα όπου υπάρχει ούτως ή άλλως μία βεβαιότητα. Ούτως ή άλλως σήμερα μπορεί κανείς μεμονωμένα να προσφύγει, αλλά δεν το κάνουν οι περισσότεροι γιατί έχουν μικρότερη δυνατότητα επιτυχίας και ακριβώς εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε το σύστημα στην ε, Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν αυτά τα συστήματα αλλά δεν λειτουργούν γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά εμπόδια από τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προσφύγουν. Γι' αυτό νομίζω έχουμε και μεγάλο βαθμό συμφωνίας και λέμε πως πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Οπότε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα μια μετριοπαθή προσέγγιση και μετά να δούμε αν μπορούμε να εξελίξουμε περαιτέρω την ε, υπόθεση, αλλά δεν σημαίνει αυτό πως ε, θα απαγορεύσουμε τις ε, μεμονωμένες ε, προσφυγές και κάτι άλλο για αυτό το οποίο είπε ο κ. Σάντς Φρεσέδο. Συμφωνώ απολύτως μαζί του. Πράγματι είναι σημαντικό το ότι ρυθμίζεται χωριστά το δίκαιο του ανταγωνισμού στην ε, συνθήκη, αλλά παρόλα αυτά η νομική βάση θα είναι το άρθρο 104 της εσωτερικής αγοράς για να έχουμε και εμείς λόγο ως συνομοθέτης. Και θα χαιρόμουν να ε, εγκριθεί αυτή η εκθέση με ευρεία πλειοψηφία και να ληφθούν υπόψη, όπως είπα, τα του δικαίου του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Θα ψηφίσουμε στις 17 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας και η έκθεση θα πάει στην Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Οπότε, σημειώνω πως ε, εξακολουθούμε βεβαίως να μην έχουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή ζώνη ώρας, οπότε είμαστε ένα-δύο λεπτάκια πίσω από την ώρα παρά τα όσα λέει το ρολόι. Καλωσορίζω λοιπόν τον Ζαν Κλου Τρισέ για το τέταρτο θέμα της ημερικής διάταξης για την δημόσια ακρόαση. Ε, καθώς καλωσορίζουμε τον Ζαν Κλοντ υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Κάτι το σχετικά νέο σε σύγκριση με τον νομισματικό διάλογο ε, καθώς μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε πάει στο νομισματικό αυτό διάλογο 35 φορέ. Οπότε, παρακαλώ όσοι ε, θέλουν να θέσουν ερωτήσεις να θυμούνται πως δεν βρισκόμαστε στο νομισματικό διάλογο. Είναι μια ακρόαση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και ανάλογε πρέπει να είναι και οι ερωτήσει. Θα δώσω τον λόγο συνήθω στον ε, πρόεδρο, στον κύριο Τρισέ για να μας κάνει μια δεκάλεπτη σύνοψη των όσων έχει να πει και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά αξιόλου στα μέλη, έχουμε πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ενώπιον σα υπό την ιδιότητά μου, όπω είπατε, κυρία Πρόεδρε, ω πρόεδρο του Συμβουλίου Συντηρικού Κινδύνου, για να σα εξηγήσω τι έχει κάνει το Συμβούλιο αυτό στο πρώτο εννεάμινο των δραστηριοτήτων του. Θα περιγράψω καταρχάς την τρέχουσα κατάσταση και την έκκληση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον συστημικό κίνδυνο για να υπάρξει δράση χωρίς καθυστέρηση. Θα παρουσιάσω στην παρουσίαση των πρώτων ε, προτάσεων που υποβλήθηκαν από το Συμβούλιο αυτό που θα δημοσιευτούν και θα κοινοποιηθούν σήμερα. Επιπλέον, κάποιες ε, μακροοικονομικές επιπτώσεις θα αναφέρω όσον αφορά τη σημερινή νομοθεσία όπου το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης έχει αρμοδιότητες και συμμετέχει. Και έτσι θα ολοκληρώσω τις, ε, την παρέμβασή μου με κάποιες παρατηρήσεις για τις τρέχουσες εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής όσον αφορά διαρθρωτικές ε, διαφορετικά μεσοπρόθεσμα θέματα. Ας ξεκινήσω περιγράφοντας τη σημερινή κατάσταση πως έχει και τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν όπως πιστεύουμε εμείς. Η κρίση αυτή έφτασε μια συστημική διάσταση πλέον που έχει λάβει. Όπως είπε το Συμβούλιο σε συνέντευξη τύπου, σε δήλωση προς τον τύπο, αμέσως μετά την γενική συνάντηση του Συμβουλίου στην 21η Σεπτεμβρίου πέρυσι, η πίεση από τις μικρότερες ε, οικονομίες ε, μετακινήθηκε σε μεγαλύτερες χώρες. Είναι προφανής η ένταση αυτή όσον αφορά τα ομόλογα, ενώ η ευμεταβλητότητα των αγορών δείχνει ότι οι εντάσεις έχουν διαχυθεί και έχουν διαδοθεί στις κεφαλαϊκές αγορές παγκόσμια. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση από το στέγνομα των κεφαλαίων από πλευράς τραπεζών η αλληλοσύνδεση όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα οδήγησε σε αυξανόμενο κίνδυνο όσον αφορά την επιμόλυνση και διάδοση αυτού του φαινομένου. Όσον αφορά τη σταθερότητα, έχει ε, υπονομευθεί όσον αφορά την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η κατάσταση συνέχισε να είναι πολύ απαιτητική και έντονη. Είναι συστημική η κρίση αυτή και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος αποφασιστικά. Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι εθνικές ε, κρατικές αρχές καθώς επίσης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να δράσουν από κοινού ταχύτατα. Περαιτέρω καθυστερήσεις μόνο συνεισφέρουν στο να επιδεινωθεί ακόμα περαιτέρω η κατάσταση. Στο άμεσο μέλλον υπό το πρίσμα του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου τα μέτρα αυτά τα οποία για τον, ε, τον χώρο της Ευρωζώνης που είχαν συμφωνηθεί την 21η Ιουλίου πρέπει πλήρως να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν και με ταχύτητα. Αξιόπιστη και αηφόρα δημοσιονομική πολιτική με τη διάρθρωση των, ε, με διεύρυνση των διαθωτικών μέτρων πρέπει να επιτευχθεί ώστε να διαφυλαχθεί και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των εμπλεκόμενων στις παγκόσμιες αγορές. Συντονισμός και συνέπεια πρέπει να διευρυνθούν και τονίζω για άλλη μια φορά ότι είναι θέμα κατεπήγον αυτό. Πρέπει όλοι να δράσουν, όλες οι αρχές να δράσουν ευθυγραμμιζόμενες και συντονιζόμενες ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα. Πρέπει να συντονιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών με, χρησιμοποιώντας ε, τις διευκολύνσεις και τα μέσα στη διάθεσή τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει διαφανής αξιολόγηση όσον αφορά την έκθεση σε κινδύνους το μέσο για την διευκόλυνση αυτή θα πρέπει από πλευρά των κυβερνήσεων να χρησιμοποιηθεί για την α, ε, επανακεφαλαίωση των τραπεζών και αυτό θα μπορούσε να είναι υποφελές. Τώρα θα ήθελα να αναφέρω κάτι άλλο, τις συστάσεις για δανεισμό σε ξένο συνάλλαγμα. Σήμερα η ESRB δημοσιεύει τις πρώτες συστάσεις της από πλευράς της ε, για τον δανεισμό σε ξένο συνάλλαγμα, σε ξένα νομίσματα. Και Τώρα όταν δημοσιεύεται, δεν δημοσιοποιείται, παρουσιάζεται έτσι και στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει να δούμε την έκθεση στον κίνδυνο αυτών των ε, συναλλαγμάτων αυτών, στον οποίο εκτίθενται τα κράτη και είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους ε, για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Να αναφερθώ στους τρεις κυριότερους κινδύνους που υφίστανται. Πρώτον, με την έκθεση των δανειστών όπως των οικοκυριών στους κινδύνους των ξένων αυτών συναλλαγμάτων. Εδώ υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου ε, το οποίο ο θα ε, έπρεπε να μας κάνει να δούμε ότι αυξάνεται πολλές φορές ε, η αξία του δανείου που πρέπει να αποπληρωθεί. Επίσης, σε σχέση με τέτοια δάνεια μπορούν να συνεισφέρουν σε υπερβολικά επίπεδα δανεισμού. Επίσης ε, έχουμε λόγω της υπερβολικής εξάρτησης ε, από βραχυπρόθεσμες ε, τέτοιες αγορές κινδύνους. Μια και υπάρχουν κίνδυνοι για την ε, δημοσιονομική σταθερότητα, ο κίνδυνος διασυνοριακής μόλυνσης ή διάχυσης του κινδύνου πρέπει να δώσει δυνατότητα να δράσουμε άμεσα. Αποφασίσαμε να συντάξουμε συστάσεις για την πολιτική. Αυτές οι συστάσεις επικεντρώνονται στις πολιτικές δράσεις για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από νέα δάνεια όσον αφορά δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα προς τους ε, δανειστές. Επιπλέον οι συστάσεις ε, που παρουσιάζουμε σήμερα στοχεύουν στο να δώσουν μια πλήρη απάντηση πολιτικά σε σχέση με την υπερβολη, τον υπερβολικό δανεισμό όσον αφορά ξένα νομίσματα. Θα πρέπει να δούμε εδώ την ε, αντοχή και την ε, ενδυνάμωση της αντοχής ε, του ε, χρηματοοικονομικού τομέα που πρέπει να πετύχουμε. Ας ανακεφαλαιώσουμε και να δούμε αυτές τις συστάσεις χωρίς να επισέλθουμε σε υπερβολικά σε τεχνικές λεπτομέρειες. Πρώτον, συνιστούμε να ζητηθεί από τις αρχές τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να δίνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των δανειστών για τους κινδύνους και να αυξηθεί η αξιοπιστία σε σχέση με το πλαίσιο δανεισμού για νέους δανει, ε, δανειζόμενους που προσφεύγουν σε αυτό το μέσο. Επίσης πρέπει να αποφευθεί υπερβολική, ε, υπερβολικό εύρος τέτοιου δανεισμού και να βρεθούν τα μέτρα να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος. Τρίτον, συνιστούμε να ζητηθούν από τις αρχές από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να ληφθούν πλήρως υπόψη οι κίνδυνοι στο εσωτερικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων από πλευρά τους και να υπάρχει επαρκές κεφάλαιο για την κάλυψη τέτοιων κινδύνων. Και τέταρτον, συνιστούμε οι αρχές να επαγρυπνούν όσον αφορά τέτοιους κινδύνους και να εξετάσουν τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών όπου αυτό καταστεί αναγκαίο για τις ε, αρχές αυτές ε, η δημοσιοποίηση αυτών των συστάσεων καθορίζει την έναρξη της φάσης ε, εφαρμογής και υλοποίησης και για το ESRB θα είναι η αρχή, η έναρξη της περίοδου εποπτείας. Με βάση το μηχανισμό αυτό οι αρχές θα έχουν προθεσμία μέχρι το 2012 ή 2013. Αυτό θα εξαρτάται από τις ατομικές συστάσεις προς αυτές για να υλοποιήσουν, να δράσουν και να υλοποιήσουν αυτές τις συστάσεις πλήρως. Η ESRB θα αξιολογήσει μετά αυτές τις δράσεις ή σε περίπτωση μη ανάληψης ε, δράσης ε, θα εξετάσει τις δικαιολογίες ή τα επιχειρήματα και θα αποφασίσει για τη συνέχεια που θα δοθεί από πλευρά τη. Όπως γνωρίζετε το ESRB θα αναφέρεται πάντα στο Ευρωκοινοβούλιο σε περιπτώσεις ε, όπου θα θεωρείται ανεπαρκής η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Και σας διασφαλίζουμε ότι είναι σαφέστατο ότι εμείς ε, θα το κάνουμε αυτό όπως ε, πρέπει και όπως χρειάζεται. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να σας πούμε ότι ε, αντιμετωπίζοντας ε, την ευμετάβλητη κατάσταση και τον ευάλωτο χαρακτήρα αυτού του δανεισμού, η SRB ε, εξετάζει συστημικούς κινδύνους που θα μπορούν να προέρχονται από δανεισμό όσον αφορά τις τράπεζες σε ξένα νομίσματα, σε ξένο συνάλλαγμα. Εξετάζεται άμεσα η δυνατότητα ανάληψης δράσης ε, για να αντιμετωπιστεί ο ευάλωτος αυτός χαρακτήρας όσον αφορά ε, τον δανεισμό αυτό η ε, προηγούμενη εργασία, το προηγούμενο έργο έχει βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν οι αρχές το συστημικό κίνδυνο που προέρχεται από την υπερβολική εξάρτηση από χρηματοδότηση σε δολάρια για παράδειγμα. Έτσι πρωτογενώς θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω η δυνατότητα αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων και να ενισχυθούν τα προγράμματα των τραπεζών για την επαρκή χρηματοδότησή τους. Η SRB θέλει να αποφύγει την μελλοντική επανάληψη αυτών των περιπτώσεων που είχαμε βιώσει στο παρελθόν το 2008 και το 2011 και που μπόρεσαν να ρυθμιστούν μέσω των πολυμερών συμφωνιών, μέσω των μεγαλύτερων τραπεζών. Επιτρέψτε μου να στραφώ τώρα σε κάποιες νομοθετικές προτάσεις επί των οποίων το Ευρωκοινοβούλιο είχε εργαστεί ως συνομοθέτης. Ε, τους ε, τελευταίους μήνες ως ε, Ευρωπαίοι νομίζω πως είναι σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη η οποία θα ξεκινήσει την διαδικασία εφαρμογής τη Συμφωνίας ε, Βασιλεία 3 όπως ε, εγκρίθηκε από τους ε, G20 και βεβαίως ως πρώτη η οποία θα προβεί σε αυτή την κίνηση πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει πλήρως και συνεπώς την Συμφωνία Βασιλεία 3. Οι εξαιρετικές συνθήκες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζουν την σημασία που έχει η έγκαιρη και συνεπής δράση για να αντιμετωπιστεί ο συστημικός κίνδυνος. Γι' αυτό το Συμβούλιο μας τονίζει πως οι εθνικές μακροπολιτικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ε, πιο αυστηρές συνθήκες όσον αφορά τα προληπτικά μέσα πάντα βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη τι ε, τοπικέ οικονομικέ συνθήκε. Δεν θα μα δικαιολογήσουν οι πολίτε μα εάν δεν ε, αντιμετωπίσουμε του σοβαρού συστημικού κινδύνου και ε, έχουμε βλάβη στην οικονομία γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οι αρχές να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο. Βεβαίω. δεν χρειάζεται να πω πω αυτό θα πρέπει να γίνει χωρί να διακυβευτεί η ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι εύκολο. Η χρήση μακροπροληπτικών εξουσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί και πρέπει να συμφιλειωθεί με την μη παραβίαση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβουλίο μας, δεδομένης της έντολής του, μπορεί να αναθεωρήσει αποφάσεις που ελήφθησαν στο εθνικό επίπεδο από τις μακροπροληπτικές αρχές για να ειδοποιήσει την Κομισιόν για τυχόν παραβάσει και να φροντίσει οι εθνικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τυχόν διασυνοριακές συνέπειες. Έχοντας αυτά κατά νου, εξετάζουμε και θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε τα σχέδια κανονισμών για τις ε, τράπεζες, τον ΕΜΗΡ, τις υποδομές των αγορών, καθώς και την Οδηγία Περιφερειακότητας 2 από μια μακροπολιτική σκοπιά έτσι ώστε να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία δράσης και πάντα σύμφωνα με την εντολή μας περί μακροπροληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ε, είναι απαραίτητο θα κάνουμε συστάσεις στο Κοινοβούλιο και στους υπόλοιπους νομοθέτες για να ενισχυθούν οι μακροπροληπτικές στοιχές της σχεδιαζόμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τώρα θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την δουλειά μας η οποία συνεχίζεται σε πιο δομικά, μέσω πρόθεσμα ζητήματα, στο πλαίσιο της γενικότερης ανησυχίας η οποία υπάρχει για αγοραπολισίες υψηλής συχνότητα, ε, συχνότητας. Απαντήσαμε με κάποιες μακροβουλευτικές πρωτοβουλίες ε, από την ε, ΕΣΜΑ η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή των Χρηματαγορών. Πρώτα απ' όλα για το UCITS και τα τα μία τα οποία διαπραγματεύονται εκεί πέρα. Οι απαντήσει μας, η οποία βεβαίως είναι δημοσιευμένη μας ε, στο ενιστοσελίδα μας, διασφαλίζει πως τα μαθήματα του παρελθόντος λαμβάνονται υπόψη προληπτικά. Η πείρα μας παραδείγματος χάρη με περίπλοκα προϊόντα έχει δείξει πως η κίνδυνη σε αυτά ίσως δεν είναι πλήρως αντιληπτή και όχι μόνο από αυτούς οι ε, οποίοι είναι καταναλωτές λιανικής, αλλά ακόμα και από θεσμικούς και άλλους επενδυτές δεδομένης δε της ασάφειας και της περιπλοκότητας αυτών των προϊόντων, όπως παραδείγματο χάρη τα συνθετικά ETF, το Συμβούλιο μας προτείνει να εξετάσουμε την δυνατότητα απόσυρσης του σήματος UCITS από τέτοιες δομές για να παραμείνουν τα προϊόντα απλά και έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη στο σήμα της ε, UCITS εάν, τα προϊόντα αυτά έχουν προβλήματα στο μέλλον. Δεύτερον, για τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας αναγνωρίζουμε πως η τεχνολογική πρόοδος έχει συνεισφέρει στην δυνατότητα των αγορών στο να παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην πραγματική οικονομία. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία έχει δείξει πως η χρηματοπιστωτική καινοτομία συχνά εμπεριέχει τον κίνδυνο συστημικού κινδύνου, οπότε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές θα πρέπει να γίνονται πλήρως αντιληπτές και να παρακολουθούνται προσεκτικά. Πρέπει άρα να ερευνήσουμε περαιτέρω τον πιθανό βλαπτικό ρόλο των συναλλαγών αυτών στη ρευστότητα και το πώς πιθανώς μπορούν να ενισχύσουν τα σοκ των αγορών. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την εποπτεία μας αλγοριθμικών συναλλαγών και να προτείνουμε μέτρα πιο προληπτικής φύσης, παραδείγματος χάρη εργαλεία διαχείρισης κρίσεων και διαρθρωτικά μέσα τα οποία αξίζουν περαιτέρω μελέτης. Θα ήθελα τώρα να ολοκληρώσω την παρουσίαση του έργου της, ε, του Συμβουλίου μας τους πρώτους μήνες της ύπαρξής του. Είμαι περήφανο για το ότι είμαι ο πρώτος ε, πρόεδρος του Συμβουλίου αυτή μαζί με τον, Συμβουλίου μαζί με τον Μέρβιν Κίνγκ και τον ε, Ανδρέα Ανδρέα. ξέρω πως το Συμβούλιο σας είναι ιδιαίτερα αγαπητό γιατί αποφασίσετε εσείς να το δημιουργήσετε. Εύχομαι λοιπόν στον διαδοχό μου τον Μάριο Ντράγκη καλή επιτυχία και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 Σημαντικό να ληφθούν σαφείς αποφάσεις οι οποίες θα είναι στο ύψος και στην σοβαρότητα της κατάστασης. Ε, ε, Σε ό,τι αφορά τώρα την τράπεζα Dexia, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, παρά μόνο ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και στις δύο ή μάλλον τρεις χώρες ε, οι οποίες πλήττονται, όλες οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί να εφαρμοστούν άμεσα Πιστεύω ότι αυτές οι αποφάσεις είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο δύο πόλμα. Ένα λεπτό. Ας Άστονε, κύριε Πρόεδρε. Για τον επιφυλακτικό τρόπο έκφρασή σας παρόλα αυτά με εξαιρετικά σαφή τρόπο επισημάνατε Πρόεδρε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση και περίοδο στην Ευρωζώνη. Η κοινοβουλευτική μα ομάδα εδώ και 1,5 χρόνο έκρουε κόδωνα κινδύνου τα κράτη-μέλη να μην καθυστερήσουν στην αντίδρασή τους. Δεν είναι τώρα η χρονική στιγμή επιτέλους να κινητοποιηθεί ταχύτερα το ESFS και δεν είναι τώρα η ώρα να δώσετε άδεια λειτουργίας στο ESFS ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει έγκαιρα, νωρίς ώστε να μπορέσουν τα πράγματα να καταλήξουν στην ορθή κατεύθυνση. Η κεφαλοποίηση όσον αφορά τα κράτη-μέλη και πάλι δείχνουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να καλυφθούν. Όμως η υπερχρέωση των κρατών μελών εκ νέου θα επιβαρυνθεί. Πείτε μας γιατί ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου δεν είναι υπέρ του να δοθεί αυτή η άδεια λειτουργίας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσον κατάλαβα το ερώτημά σας. Δεν είμαι υπέρ της έκδοσης τραπεζικών αδειών. Όχι, νομίζω εννοήσατε την ε, λειτουργία του στηρητικού προσωρινού μηχανισμού, του EFSF. Αυτό είναι το οποίο μπορεί να υποφέρει να θέλετε, κάποια σχετική και να προσφέρει μόχλευση. Α, ναι, κατάλαβα, συγγνώμη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει πολλά πράγματα. Το ερώτημά σας όμως απευθύνεται, από ό,τι κατάλαβα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι του δικού μας Συμβουλίου, γιατί είναι σαφές. Αυτό το οποίο ζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι ο μηχανισμός να είναι στο δυνατόν πιο ευέλικτος και πιο ανοιχτός και να εφαρμοστεί στο δυνατόν νωρίτερα και με την κατάλληλη μόχλευση. Ε, αυτό το οποίο μετράει το δικό μας Συμβούλιο είναι η μόχλευση που εξαρτάται εν πολλής ε, από την βούληση κάθε κυβέρνηση να μοχλεύσει από τον προσωρινό μηχανισμό, το EFSF, θα είναι όσο το δυνατόν ανάλογο στη σοβαρότητα τη κατάσταση. Αυτό είναι σαφέ. Εάν έχετε ερώτημα τώρα για το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι άλλον έκδοτο. Δεν έχω την άδεια να απαντήσω με άλλη ιδιότητα εδώ. Μου τη δίνετε? Ωραία. Λοιπόν, έχω τώρα την ιδιότητα του Διευθύνοντο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπω ξέρετε, το σχετικό Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει πάρα πολλέ σημαντικέ αποφάσει και ξέρετε καλύτερα από του περισσότερου ότι κάποιε από τι αποφάσει αυτέ όλε στοχεύουν στην, στο να επιτραπεί καλύτερη αποκατάσταση τη ε, παρακολούθηση των νομισματική πολιτική μα και θεωρούμε ότι είναι πολύ τολμηρέ οι αποφάσει που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένη και τη παρέμβαση στην δευτερογενή αγορά. Θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει έχουν κάθε δυνατότητα να μοχλεύσουν από μόνε τους τον μηχανισμό, τον EFSF, με τι κατάλληλε αποφάσει που πρέπει να λάβουν. Και δεν θεωρούμε ότι θα ήταν πρόσφορο για μα να κάνουμε μόχλευση του μηχανισμού αυτού. Είναι τη ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυβερνήσεων και των Κεντρικών Τραπεζών των Εθνικών και έχουν κάθε τρόπο και όλα τα μέσα για να το πράξουν. Ευχαριστούμε, ε, κύριε Σιλβί. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ήμουν ε, η μετριόφρον συντάκτρια τη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για του Συστημικό κίνδυνο. Δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόσασταν τόσο γρήγορα να έρθω εδώ και να μα πείτε ότι όντω βρισκόμαστε εν το μέσο συστημικού κινδύνου. Αλλά ίσω αποδεικνύει ότι δεν δουλέψαμε το τίποτα και δεν ανησυχούσαμε ανεφλόγου. Έχω ένα ερώτημα να σα θέσω, μπορεί να μην απαντήσετε ίσω. Αλλά όπω είπατε πολύ σωστά, 21 <coughs> Σεπτεμβρίου υπήρξε μια συνάντηση. Είπατε κάποια πράγματα Εκτιμώ ιδιαίτερα το οποίο ήρθατε με τα παρησίες να το πείτε εδώ σήμερα. Ποια είναι η όλη σας αίσθηση σε ό,τι αφορά την αντίδραση των κρατών μελών. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάλι αν θέλετε να διαχωρίσετε τις δύο ιδιότητες μεταξύ των δύο προεδριών που έχετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς για να μεταφέρουμε κάποιο μήνυμα. Γιατί θυμάστε την επιμονή με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να σα τοποθετήσει στην, ε, στο φόκο αυτό τη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Ήταν και τα μηνύματα που πέρασαν για να υπάρξει και να ε, κρουστεί ο του κινδύνου, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Κοιτάξτε, ενεργοποιήσαμε με όλους τους δυνατούς διάβλους το μήνυμά μας, ζητώντα από το σύνολο των θεσμικών οργάνων και προφανώς από τις εκτελεστικές εξουσίες των κρατών μελών να λάβουν όλα τα ανάλογα μέτρα, σε μια κατάσταση την οποία χαρακτηρίζουμε εξαιρετικά σοβαρή, εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα όπως ξέρετε, και την οποία χαρακτηρίζουμε σωστημικού κινδύνου με σαφέστατο τρόπο. Ενεργοποιήσαμε λοιπόν όλα τους δυνατούς διάβλους επικοινωνίας με τις κυβερνήσεις, ώστε να τους ζητήσουμε να δράσουν με υπεύθυνο, ταχύτατο και ολοκληρωμένο τρόπο στο ύψο των περιστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, που είναι ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρόκληση, γιατί βρισκόμαστε στο επίκεντρο μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αυτού λεχθέντο λοιπόν θα αποφανθώ μετά τις συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί, έχοντας επίγνωση ότι έχουμε μείζωνα προβλήματα. Το ένα είναι του χειρισμού του, του κινδύνου των εθνικών ε, κρατών που βλέπουμε να αναπτύσσονται ταχύτατα και που ζητά να είμαστε και πάνω, αν θέλετε, και κυρίαρχοι της κατάστασης, το οποίο δεν συνέβη μέχρι στιγμής, και εξάλλου έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μία κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που επίσης και αυτή ζητά κατάλληλη απάντηση. Και οι δύο καταστάσεις ζητούν την κατάλληλη και την ταχύτερη δυνατή απάντηση. θεωρώ ότι το σύνολο του νομοθετικού έργου που ζητήσατε και που εκπονήσατε είναι χρήσιμο υπό τις περιστάσεις όπως αυτές τις οποίες βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα διαθέσιμου τους διαθέσιμους διάβλους επικοινωνίας που έχουν ε, στην, στα πλαίσια της δευτερογενούς ε, νομοθέτησης. Σας ευχαριστώ για τους ε, Ευρωπαίους Συντηρητικούς Σας ευχαριστώ. Προς έκπληξη πολλών ε, Βέλγων, ε, η Τράπεζα Δεξιά, ειδικά ο βελγικός ε, τομέας, είχε ήδη εθνικοποιηθεί από μια χώρα η οποία ήδη έχει μεγάλα βάρη. Μετά από δύο stress test λοιπόν υποφέρεται από παρεστήσεις ε, κύριε Τρισέ. Πώς ε, βλέπετε λοιπόν την επίπτωση της τραπεζικής κρίσης στο δημόσιο χρέος γιατί θα υποβεβαστεί ξανά το Βέλγιο και η Γαλλία μάλλον θα χάσει την αξιολόγηση 3α. Οπότε μία ε, χώρα ξυλώνει μία τράπεζα, αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίστροφα. Και τέλος θα ε, ήθελα να σα υπενθυμίσω τον πρώην συναδελφό σα, τον κύριο Γκρίνσπαν, ο οποίο βγήκε σύνταξη και θεωρούταν ήρωα και μετά ε, από ένα χρόνο μόλις θεωρήθηκε άρχον της καταστροφής. Οπότε και εσείς τώρα που ακούτε τους επένους χαρείτε τους γιατί μπορεί να μην κρατήσουν και πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να πω πως προειδοποιώ τις κυβερνήσεις και όλες τις ε, υπεύθυνε ε, αρχές, τις προειδοποιούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποτέ δεν είχαμε επαναπαυθεί είτε υπό την ιδιότητα του, εγώ προσωπικά, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας. Ποτέ δεν είχα επαναπαυθεί. Και πριν από λίγε ημέρες επανέλαβα πως στην πρώτη μου ακρόαση ενώπιον του Κοινοβουλίου είπα πως το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη έχει κέρια σημασία. Δημοσιονομική, η δημοσιονομική συνέπεια έχει κέρια σημασία. Αυτά μόνο να αναφέρω και πολλές άλλες προειδοποιήσεις ε, τις οποίες είχαμε απευθύνει και βεβαίως μιλούσα ε, εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο από την άλλη. Οπότε Καθόλου δεν είχαμε καθυσυχάσει. Μου ασκούσαν κριτική μάλιστα οι κυβερνήσει και μου λέγανε πω δραματοποιείται τα πράγματα, δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση κτλ. Και κάποιοι ε, βουλευτέ ε, από διάφορε χώρε νομίζω μπορούν να το βεβαιώσουν. Οπότε ποτέ δεν υπήρχε ευσυχασμό. Αλλά τούτου λεχθέντο βεβαίω υπήρχαν κάποια ζητήματα σημαντικά και όταν κρύγνεται προβλήματα από εδώ και από εκεί, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα. Κάτι το οποίο γίνεται τώρα και για την τράπεζα που αναφέρατε. Ε, ζήτησα από όλους τους ε, εταίρους και τις αρχές να το κάνουν γρήγορα, αποτελεσματικά, γιατί πάντα ο χρόνος μετράει όταν υπάρχουν μεγάλες ε, δυσκολίες και ε, αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ε, εδώ πέρα πρέπει να πούμε πως ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας ειδικά στήριξε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αντιστάθηκε σε πιέσεις από τα κράτη-μέλη και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το ρόλο γιατί η ανεξαρτησία της ε, τράπεζας και οι δράσεις ε, τις οποίες ε, έλαβε νομίζω ήταν σημαντικές. Κατόπιν η πράσινη, ο Σβέν. Κύριε Τρισέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω πως σήμερα μάθαμε γιατί δημιουργήσαμε αυτό το θεσμικό όργανο. Καλώς ορίζω πολλές από τις λεπτομερείς συστάσεις σας, ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε για το usage θα πρέπει πράγματι να, να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία είπατε. Έχω ένα πιο γενικό ερώτημα. Η οικονομία εξακολουθεί να είναι υπερβολικά μοχλευμένη. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος σε σχέση με την πραγματική οικονομία. Και βεβαίως ε, ο πληθωρισμός ε, έχει αποκλειστεί από τις συνθήκες ως μέσο περιορισμού αυτής της μόχλευσης. Οπότε ποια άλλα μέσα προτείνεται για την απομόχλευση του χρηματοοικονομικού τομέα προς όφελος πραγματικής οικονομίας. Τι ορίτε για έναν ευρωπαϊκό φόρο επί του πλούτου για να μειωθεί το δημόσιο χρέος και να μειωθεί η μόχλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ αυτά που είπατε για τα τεχνικά θέματα και θεωρούμε πραγματικά ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή συναγερμό όσον αφορά τα νέα τεχνολογικά μέτρα και μέσα όσον αφορά για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Και πάλι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε στο ύψος των περιστάσεων αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων όσον αφορά την τεχνολογία καινοτομία και όσον αφορά και τον ευφύ τρόπο δράσης. Για το ερώτημά σας, πρώτον δεν θα τοποθετηθώ ε, αντικειμενικά για την απόφαση που πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις για το πώ εκείνε θέλουν να διοργανώσουν θέματα φορολογίας και φορολόγηση και για την δική σας πρόταση για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό για την φορολόγηση του πλούτου από τις κυβερνήσεις ε, στα δημοκρατικά καθεστώτα μας ε, πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί αυτό. Βλέπουμε όμως μετά από μια μεγάλη περίοδο μόχλευσης παγκόσμια, μια περίοδο επανόρθωσης ή διορθωτικών κινήσεων και γι' αυτό πάντα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί και συνετοί γίνεται γιατί σε περίοδο ασύνετης δράσης υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα και διαταράξεις. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ευρώπη θα έλεγα είναι ότι οι χρηματοδοτούνται από τα, τον χρηματοοικονομικό τομέα οι οικονομίες μας σε 75% όταν σας είπα το ποσοστό είναι 25% όπου οι αγορές χρηματοδοτούν 75% της οικονομίας ενώ σε αυτή την πλευρά στην Ευρώπη δηλαδή είναι 25% η χρηματοδότηση μόνο από τι αγορέ. Γι' αυτό οι ισολογισμοί των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι τόσο σημαντική υπόθεση. Και τι λέμε, λέμε ότι για να καταφέρουμε να αποφύγουμε ακριβώ αυτή την απομόχλευση που είναι, θα ήταν κάτι το αναπόφευκτο. Δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε ε, παρέμβαση αρνητικά στην ε, ε, χρηματοδότηση της οικονομίας και θα πρέπει να κεφαλοποιηθούν περισσότερο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ώστε να μην υπάρξει συρρήκνωση των ε, ισολογισμών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε τη πραγματική οικονομία. Και αυτό πραγματικά, όπω και πρόσφατα αναφέρθηκε, θα πρέπει να, μπορέσει, να, να μπορέσουν να είναι υγιεί ε, οι ισολογισμοί του, ώστε να μπορούν σε σχέση με την ε, διαδικασία χρηματοδότηση των πακέτων ακριβώ όσον αφορά και τις ε, την αντιστάθμιση, να υπάρξει και η σωστή επανακεφαλοποίηση, πράγμα που χρειάζεται όπου χρειάζεται στο επίπεδο της Ευρώπης συνολικά, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα σημαίνει είτε ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να επανακεφαλοποιηθεί ο ίδιος για να αντιμετωπιστούν οι στενοποί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να προστατευτεί η πραγματική οικονομία όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα. Ευχαριστώ ομολογώ ότι είμαι ανησυχήση. Αν θέλουμε να μειώσουμε το χρέο, πρέπει από την άλλη πλευρά να μιλήσουμε για τη μείωση του πλούτου. Αυτέ είναι οι δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ρόλο να αποφανθεί τη φορολογία. Όταν μιλάτε ω επικεφαλή ε, του Συμβουλίου όμω, έχετε και την πλήρη εντολή και εξουσιοδότηση να μιλήσετε και για φορολογική πολιτική. Δεν περιορίζεστε από κάποιο κανονισμό υπό αυτή την έννοια. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε το βασικό ερώτημα το οποίο έθεσα. Ε, και πάλι, νομίζω ότι αυτή είναι απόφαση που πρέπει να ληφθεί από τις δημοκρατίες μας. Το να μειωθεί το ίδιο εθνικό κρατικό χρέος, αυτό μπορεί να βρεθεί είτε με την αύξηση φορολογίας είτε με την μείωση των δαπανών. Και αυτό είναι πολύ συξαρτάται από τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δημόσιες δαπάνες που είναι το 35% του ΑΕΠ και άλλες χώρες που έχουν δημόσιες δαπάνες που ξεπερνά το 55% του ΑΕΠ. Η διαφορά μεταξύ των δύο όντα δηλαδή ένα 20%. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν οι αποφάσει, λαμβάνοντα υπόψη τη συνολική κατάσταση των διαφόρων χωρών. Νομίζω ότι είναι προφανώ πολύ σημαντικό αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ξέρω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα να γίνει ανοιχτή συζήτηση, αλλά θα πρέπει να πάμε συντονιστέ. Λυπάμαι. Λυπάμαι, όχι. Ένα λεπτό, κύριε Σέντρισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μπαίνω κατευθείαν στην ερώτηση αγενός, διότι δεν υπάρχουν χρόνια για να πούμε ευγενικά λόγια. Έχω μπροστά μου τον πίνακα των spreads, των CDS, των ελληνικών ομολόγων από το site του Bloomberg. Αυτός ο πίνακας δείχνει πως τον Οκτώβριο του 2009 αυτά τα spreads ήταν λίγο πάνω από τις 100 μονάδες βάσης. Σήμερα, ένα χρόνο και κάτι μετά την έλευση της Τρόικα, την εφαρμογή του μνημονίου, εκτός από τα προβλήματα ύφεση και ανεργίας, τα spreads, κύριε Πρόεδρε, από τις 100 μονάδες βάσης του Οκτωβρίου έχουν φτάσει στις 3.500 μονάδες βάσης των CDS. Σας ερωτώ λοιπόν, αυτό σημαίνει επειδή μεταδίδεται ο ιός της κρίσης ότι έχουμε μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πολιτικές έχουν αποτύχει. Κυρία Πρόεδρε, τελείωσε. Όπως ξέρετε, έχουμε δύο σοβαρά το ένα είναι πως κάποιες χώρες ε, συμπεριφέρθηκαν με λάθος τρόπο στο παρελθόν. Και ξέρετε καλύτερα από τον καθένα πως η Ελλάδα είναι η χώρα, εάν μου επιτρέπετε, η οποία δεν συμπεριφέρθηκε σωστά στο παρελθόν, από όταν μπήκε στο ευρώ, ξεχνώντας εντελώς πως ε, το ευρώ είναι μια ζώνη όπου υπάρχει σταθερότητα τιμών, όπου είχε οικοδομηθεί για να υπάρχει σταθερότητα τιμών και όπου το βασικό μέτρο ήταν πως ο πληθωρισμός συνολικός θα ήταν 2, κοντά στο 2%. Και ελήφθησαν αποφάσεις ξεχνώντας αυτό το πράγμα εντελώς και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Αυτό έχει βασική σημασία. Πρέπει να ε, γίνει αυτή η διόρθωση και υποθέτω πως ε, γίνεται με την βοήθεια των όρων που έχει θέσει το Διεθνές ομοσπονδιακό Ταμείο και η Ευρώπη. Έτσι θα γίνει αυτή η διόρθωση. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουμε το ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση όσον αφορά το δημόσιο χρέος και αυτό υπάρχει και εκτός Ευρωζώνης, εκτός Ευρώπης, ακόμα και αν δούμε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και βεβαίως εκεί πέρα συλλογικά ως σώμα μιλάω για τα μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 17 και οι 27, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συστημική κρίση που είναι παγκόσμιας φύσης και της οποίας είστε το επίκεντρο. Είναι πράγματι ε, κάτι το οποίο για το οποίο ζητάμε μία επαρκή απάντηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε απολύτω συνεπεί στα μηνύματα που στέλνουμε ω προ αυτό. Σα ευχαριστώ. Thank very much. Uh, now... πολύ. Και τώρα εκ του ΕΛΚ. Για ένα λεπτό, Ο κύριο Λάγκαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω που αφορά το πρώτο σκέλος ε, του προλαλήσαντος στην ερώτησή του για την αξιολόγηση των κινδύνων. Έχουμε τη Βασιλεία 2 και τη Βασιλεία 3 τα ίδια κεφάλαια όσον αφορά την, ε, τα κρατικά ομόλογα και έχουμε ένα μηδενικό ε, ποσοστό. Εδώ κύριε Πρόεδρε θεωρείτε ότι αυτό είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα δεύτερον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες που έχουν προβλήματα στους ε, ισολογισμούς τους είναι πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από ότι το κοινωνικό, το ΑΕΠ των κρατών που έχουν ε, την υπερχρέωση. Θυμούμε τον πρώτο γύρο για την τέξια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο πλαίσιο 24 ωρών ενέκρινε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, χωρίς με οποιοδήποτε τρόπο να υπάρχει απέτηση για βαθιά αναδιάρθρωση ήταν τότε η υπεύθυνη για τον ανταγωνισμό επίτροπος της Ολλανδίας αρμόδια. Εδώ υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια που βλέπω. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα καταφέρει ο χρηματοοικονομικός τομέας, οι τράπεζες να, φτάσουν, να φτάσουν περισσότερο κοντά στην ε, πραγματική οικονομία χωρίς να υπάρξει συρρήκνωση. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ε, Ευχαριστώ. Στο πρώτο σας ερώτημα που υπογραμμίζει ένα από τα κύρια παγκόσμια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Η υπόθεση εργασία μέχρι πρόσφατα ήταν ότι έχουμε κινδύνους του ιδιωτικού τομέα και έχουμε το πεδίο εκτός κινδύνου που είναι, αν θέλετε, της κρατικής φύσης. Και ο λόγος για τον οποίο στη Βασιλεία 2 και Βασιλεία 3 έχουμε αυτή την υπόθεση εργασία όντως είναι ότι υπάρχουν, αν θέλετε, τα κεντρικά, αν θέλετε, ευρωφυλάκια των κρατών. Το επεισόδιο τώρα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμια κρίση και επανέρχομαι στο ερώτημα το οποίο ετέθη στο κατά πόσον είχαμε φυσικάσει ή όχι. Καθόλου δεν είχαμε φυσικάσει. Ούτε σε επίπεδο Ευρώπης, ούτε σε επίπεδα. Uh, we found ourselves that... Ε, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο ήμασταν πάρα πολύ αφιλεί και υπερβολικά σίγουροι ότι ποτέ θα αμφισβητούνταν η ε, πολιτική των Υπουργείων Οικονομικών. Λέγαμε, εστέ προσεκτικοί. Δεν είναι δυνατόν ποτέ κρατική, ε, κρατικά δημοσιονομικά να είναι υπό αμφισβήτηση ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους. Και τώρα είναι πρόκληση για όλου ανεξαιρέτω. Βρισκόμαστε επίκεντρο, αλλά είναι πρόκληση για του πάντε και αποδεικνύει σε ποιο βαθμό μπορεί να αλλάξει ταχύτατα και άρδινο ο κόσμο. Γιατί, ναι, έχετε δίκιο. Οι υποθέσει εργασία Βασιλεία 2 και Βασιλεία 3 πλέον δεν είναι ε, αποδεκτέ έτσι απλά από του συμμετέχοντε στην αγορά. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Το κύριο θέμα για μα είναι πώ θα αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του, ε, κάθε κράτους. Αυτό είναι θεμελιώδες. Εάν δεν έχουμε αξιοπιστία στο κράτος, δεν έχουμε πλέον ασφαλιστική δικλίδα, εάν ενδεχομένω υπάρχει νέα πιστοτική κρίση ή νέο δράμα του, ίδιου, του είδους που βιώσαν το 2008. Και τώρα και πάλι είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε και το, το οποίο είμαστε μάρτυρες να εξελίσσεται σε, με πραγματικούς όρους και σε πραγματικό χρόνο. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας τώρα, σε ό,τι αφορά το μέγεθος των ισολογισμών του χρηματοοικονομικού τομέα και το μέγεθος του ΑΕΠ, θεωρώ προφανώς ότι έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα να τεθούν. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ε, των ε, χρηματιστηριακών προϊόντων και του χρέους σε όλα τα πεδία και με τα νοικοκυριά και με τα κράτη, δηλαδή και σε σχέση με τον δημόσιο τομέα εν γέννη. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρούμε ότι απαιτούνται πολύ περισσότερα κεφάλαια, δηλαδή περισσότερο περιουσιακά στοιχεία, θέλετε, και λιγότερο ε, χρέος στα, στους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παναφέρθηκατε. Κύριε Τρεσέ, και εγώ θέλω να επικεντρωθώ στις κεφαλαιοχικές απαιτήσει. Υιοθετήσαμε κανόνες για αμοιβέ και τα μπόνους που τα εξασφάλισαν ότι τα υψηλά μπόνους δεν θα αφισβητούσαν την κεφαλοποίηση και την επάρκεια των ε, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Δεν είδαμε να εφαρμόζεται κάτι τέτοιο. Βέβαια, νομοθέτες όπως ε, και εσείς θέλατε να παρέμβετε για να γίνει κάτι στην περίπτωση. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, θεωρείτε ότι το Συμβούλιο σα θα δει την τρέχουσα πολιτική απολαβών για να μπορέσει να υπάρχει μια περικοπή των, ε, των ε, υπερβολικών κερδών και μπόνους και συμφωνώ επίσης ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μια όροφη, αλλά ένα κατόφλι στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την εναρμόνιση. Έχετε επαρκώς γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανησυχία σε ό,τι αφορά την μέγιστη εναρμόνιση, γιατί ίσω αυτό να υποσκάπτει την ευελιξία των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις επανακεφαλαιοποιήσει και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να πλήξει σε συστημικό κίνδυνο. Κύριε Στρισέ, οφείλω να πω ότι σε ό,τι αφορά τις απολαυέ, υπήρξαμε σαφεί. όπω ξέρετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται και σε επίπεδο του χρηματοπιστωτικού ε, συμβουλίου, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και το υποστηρίζουμε από πλευρά της Ευρώπης. Το έχουμε επαναλάβει κατά επανάληψη, ότι αποτελεί τμήμα αυτό που θεωρούμε ότι έχει ήδη καθυστερήσει, αν θέλετε, και σε ό,τι αφορά την σωστή συμπεριφορά του εν λόγω τομέα, αλλά και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ισολογισμών των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αναφορικά με τη δεύτερη παρατηρήσή σας, οφείλω να πω ότι στείλαμε σχετική επιστολή που επιβεβαιώνει την θέση αυτή, που όπως ε, αναφέρατε και εσείς, με γνωστοποίηση στον πρώτο του Κοινοβουλίου και στον πρώτο της Επιτροπής σας και επιστολή της 22 Σεπτεμβρίου. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρώτησα, λέει ο Μιλήτρια. Ναι, και στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σταλεί η επιστολή αυτή με γνωστοποίηση στου επιτρόπους Μπαγνιέ και Ρεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από Κύριε Πρόεδρε, μια σειρά μια σειρά hedge funds κάνουν τη δουλειά τους ε, με τρόπο που usage θα με ενδιέφερε αν εσείς ε, όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα το εξετάσετε σε αυτές τις ιδιομορφίες τους, στις σκιές που υπάρχουν. Θα κάνετε κάτι ώστε να μην υπάρχουν μελλοντικά κίνδυνοι. Δεύτερον, το IMF e η Κριστίν Λαγκάντες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέστησε σαφές ότι η κεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι ανεπαρκής σύμφωνα με την άποψή της. Υπήρξε κραυγή στην Ευρώπη, αλλά ούτε το SFB ούτε το RAC είχαν κάνει τίποτα. Ξέρουμε εντωμεταξύ ότι η κυρία Λαγκάρντι είχε δίκιο. Ευχαριστώ. Για τον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Θα έλεγα και πάλι, είναι ένα ζήτημα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επικεντρωθήκαμε στην πρώτη μας προσπάθεια, αν επιτρέπεται η έκφραση, στο τραπεζικό σύστημα και τις απαιτήσει του συστήματος Βασιλείας 3 και των συστημικών θεσμικών οργάνων και ούτω καθεξής. Και δεν σημειώσαμε πρόοδο όσο γρήγορα απαιτείται για την αντιμετώπιση των κινδύνων του σκιώδους τραπεζικού τομέα και για τον μοχλευτικό ή μοχλικό ε, τομέα και όσον αφορά τις ιδιομορφίες και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τεράστια σπουδαιότητας να υπάρξει αυτή η εποπτεία, ο έλεγχος, ε, έλεγχος ε, και διαφάνεια ειναι παρα πολυ σημαντικο τεραστια σπουδαιότητα να υπαρξει αυτη αφορά το σκιώδη τραπεζικό τομέα. Αυτό είναι κάτι πάλι το οποίο αφορά ένα συνολικό παγκόσμιο οικουμενικό όραμα όσον αφορά και την λέσχη των 20 και εμείς εργαζόμαστε με, όσον αφορά το στιώδη τραπεζικό τομέα καθώς επίσης και κεφάλαια το, για τις αγορές σε τεχνικό επίπεδο. Σημαντική πρόοδος ε, για την ε, αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων και της συστημικής προοπτικής και ευελπιστώ ότι ο τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη χρειάζεται την επανακεφαλαιοποίηση. Είναι μέρος του μηνύματος που αποστέλουμε αυτό και είναι ένας από τους δύο τομείς όπου πιστεύουμε ότι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και να ληφθούν ταχύτητα. Προσδοκώ, προσβλέπω να ληφθούν όσο το δυνατόν γοργότερα αυτές οι αποφάσεις ε, για να κινητοποιηθούμε. Και πάλι το μήνυμά μας είναι κρυστάλ κλά στα γερμανικά, είναι κρυστάλλινο και διαφανέστατο και σε σχέση με την Κριστίν Λαγκάντ δεν έπρεπε από την πρώτη στιγμή να υποστηριχθεί όταν δήλωσε, την πρώτη στιγμή που τα δήλωσε αυτά. Δεν είχαμε συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνάντηση του Συμβουλίου. Όταν συνήθαμε, είπαμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Και αυτά τα οποία πιστεύουμε είναι σαφέστατα ω προ αυτήν την κατεύθυνση. Και πρέπει επίση να προσθέσω ότι αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάθε μήνα τα έλεγε. Έλεγε ότι πρέπει τα έσοδά σας ε, να, ε, ε, να αποταμιεύονται, να τα κρατάτε για να αντιμετωπίσετε κινδύνους και ανάγκες και αυτό είναι ακριβώς η πτυχή εκείνη που αφορά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αυτά τα οποία ε, σε σχέση με την Ευρώπη δεν ήταν μόνο η ανάγκη επανακεφαλοποίησης των τραπεζών αλλά η μεθοδολογία σε σχέση με τις ε, διαφορετικές ας το πούμε έτσι απεικονίσεις ε, των αναγκών τραπεζικά. Δεν υπήρχε όμως καμία αμφισημία αν μου επιτρέπετε σε σχέση με το μήνυμα που στείλαμε. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση από το ΕΛΚ η Ντανούτα Γεσλοβιέσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πως ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, ειδικά σε καιρούς δύσκολους. Τα θεσμικά όργανα τα οποία αποτελούν τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας άρχισαν να ενεργοποιούνται μόλις πριν από μερικούς μήνες και γνωρίζαμε πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν υπήρχε μεγάλη δραστηριοποίηση. Πώς κρίνετε λοιπόν την αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει να σας κλωνοποιήσουμε εσάς για να βρουν πιο γρήγορα αυτά τα όργανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο πως δημιουργήσατε εσείς και δικαίως μια νέα αρχή η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Εποπτεία των Τραπεζών και αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι πως η αρχή αυτή καταβάλει προσπάθεια να ανταποκριθεί στις τεράστιες ευθύνες που έχει ε, υπό τις παρούσες συνθήκες και το βλέπω αυτό γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά τόσο ο Ανδρέα Ενρία που είναι επικεφαλής αυτής της αρχής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ε, εργάζεται πάρα πολύ τραστήρια ειδικά στην κατεύθυνση που λέτε. Βεβαίω, τα πράγματα είναι περίπλοκα στην Ευρώπη. Έχουμε 27 αρχές, 27 χώρες, 27 φορολογούμενους και 27 ε, διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας. Ε, δεν απλοποιεί τα πράγματα, λέει η Ευρώπη είναι η Ευρώπη και πρέπει να δεχτούμε το θεσμικό πλαίσιο όπως είναι. Ακόμα και αν κάποιοι από θεωρούν πως πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί για τα όσα γίνονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και το σύνολο των εποπτικών αρχών ε, στις συνθήκες αυτές βεβαίως βασίζονται και στην εκτελεστική εξουσία όταν ε, πρέπει βεβαίως να κινητοποιηθούν, όπως σας είπα, αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Οπότε η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά θα έλεγα πως όλες οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν τις ε, αυτής αυτής συμπεριλαμβανομένης. Σας ευχαριστώ, Έντβαρτ Σικλούνα. Κύριε Πρόεδρε, όταν ε, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δημιουργήθηκε, είπαν πως χρειάζονταν περισσότερη έρευνα για να βρεθούν ε, τα τραπεζικά εκείνα ιδρύματα τα οποία εγκυμονούν περισσότερο κίνδυνο. Υπό το φως των ε, πρόσφατων εμπειριών, πώς ε, έχουν αλλάξει αυτά. Δηλαδή, ποιο είναι το προφίλ ενός τέτοιου ιδρύματος. Είναι εθνικό ή διεθνές. Και όσον αφορά το ΙΦΣΕΦ, ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο θα είναι πιο ευέλικτο σε σχέση με τα όσα θεωρεί το Συμβουλίο σας για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, όπως ξέρετε, έχουμε βεβαίως εστιαστεί πάρα πολύ στον ε, συστημικό κίνδυνο στο Συμβουλίο μας. Αυτό θέλατε και βεβαίως μιλάμε κυρίως για τους ε, συστημικούς ε, τα συστημικά ιδρύματα τα οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και εφαρμόζουμε στην Ευρώπη κάτι το οποίο ισχύει παγκοσμίω, γιατί ξέρετε αυτά τα εξετάζει η Επιτροπή της ε, Βασιλείας και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Οπότε στον τομέα αυτών και όπως και αλλού υπάρχουν κάποιες παγκόσμιες αρχές τις οποίες εφαρμόζουμε σε κάθε ήπειρο, σε κάθε οικονομία συστημική. Οπότε, όπως είπαμε, πρόκειται για κάτι το οποίο είναι εν εξελίξη, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά όσον αφορά δε... τα ιδρύματα τα οποία δεν είναι τράπεζες ε, και παίζουν επίσης ένα συστημικό ρόλο λόγω μεγέθους ή διασύνδεσης είναι κάτι το οποίο είναι εν Αλλά, όπως είπατε, είναι και δύσκολο. Όσον αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εμείς πάντα λέγαμε πως θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο ευέλικτο και ανάλογο με τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δεχτούμε πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει να περάσει από 17 κοινοβούλια, 17 δημοκρατίες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυτή τη βάση και το βλέπετε γιατί είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και πρέπει να περάσει, όπως είπα, από όλες αυτές τις δημοκρατικές δικασίες. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα κάτι πιο, ε, πολύ πιο ευέλικτο και δυνατό να κινηθεί επιχειρησιακά και να μην εξαρτάται από τόσες πολλές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά αυτή είναι η απόφασή μας και πρέπει να την σεβαστούμε, να σεβαστούμε τις δημοκρατίες μας και την λειτουργία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, που δεν, λίγο χρόνο που δεν λαμβάνει το ΕΛΚ. Όποιος θέλει λοιπόν ελεύθερος χρόνος για κάποιον θέλει να θέσει ερώτημα. Ζων Πολ. Ένα σύντομο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ένα σχόλιο μάλλον περισσότερο παρά ερώτημα. Είπατε προηγουμένω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα το συντομότερο δυνατό γιατί είναι μετρημένο ο χρόνο. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο και αποδείξατε ότι ξέρετε πώ να το κάνετε. Μιλήσατε όμω για τι εποπτικέ αρχέ. Από πλευρά μου είναι εξαιρετικά απογοητευμένο. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα τη ελπίδα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τρει μεγάλοι, μεγάλοι φορεί υποπτική ούτε διαπιστευμένοι, ούτε εποπτευόμενοι. Έχει δημιουργηθεί ένα προσωρινό μηχανισμό, υπάρχει μπλοκάρισμα από πλευρά ε, του κολεγίου των εποπτών και αυτό είναι καλό σήμα, κακό σήμα. Δεν λέω ότι θα άλλαζε πάρα πολλά, αλλά ο κανονισμό σε ό,τι αφορά του ε, ε, οίκου βαθμολόγηση, πιστοληπτική ακαιρεότητα, είναι ο μόνο κανόνα που πρέπει να εφαρμοστεί και ο οποίο δεν εφαρμόζεται για τις κανόνες λειτουργίας των ε, οίκων αυτών. Είπα προηγουμένως ότι και εμείς οι ίδιοι ε, ε σε διαβούλευση που γινόταν από την Ευρωπαϊκή Αρχή, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Χρηματαγορών. Δεν ε, υπονοώ βέβαια ότι δεν είναι στο ύψος των ε, ευθυνών της η αρχή αυτή και πολλοί είπατε ότι όντως ήταν εξαιρετικά σημαντική η λειτουργία και να υπογραμμίσουμε τις ε, δυνάμει δυσκολίες που συνδέονται με τις διάφορες ίσως ε, ενδεχομένως παρακινευμένες ε, καινοτομίες σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία ή τις τεχνολογίες της συναλλαγών υψηλής συχνότητας, τα high frequency trading. Όντως σημειώνω το σχολείο σας σε ό,τι αφορά την ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Χρηματαγορών και είναι σημαντικό να δούμε την κατάλληλη εφαρμογή αυτών που εφαρμόστηκαν σε ό,τι αφορά τους οίκους βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας. Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και ερχόμαστε στο πέρας της ακρόαση αυτής. Μας δώσατε κάποια πολύ σημαντικά ε, μηνύματα σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα τη κατάστασης που αντιμετωπίζουμε και κάποιες πολύ σημαντικές και σοβαρές κρυφτικές γραμμές σε ό,τι αφορά την ανάγκη εφαρμογή κάθε είδους ε, ε, μηχανισμών διάσωσης, όπως ε, του μηχανισμού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, που θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο. Συμφωνώ προσωπικά σε αυτό. Υπάρχει πολύ έντονη κριτική η οποία έχει στραφεί εναντίον των μηχανισμών αυτών αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκαν. Ευχαριστούμε. Σας δώσαμε το επίσημο χαιρετιστήριο τελευταία φορά στον ε, τελικό χρηματοοικονομικό διάλογο. Νομίζω τώρα ότι αυτή τη φορά το αντίο είναι όντω αντίο. Έχουμε ίσω ένα δεκαπενθήμερο ακόμα στη διάθεσή μα που ενδεχομένω ξαναπροσκαλέσουμε αν συμβεί κάτι έκτακτο. Ελπίζουμε να μην συμβεί. Πάντω, τι θερμότερε ευχέ μα και όπω ακούσατε και πριν, δεν θέλουμε πραγματικά να εξαφανιστείτε με την σοφία σας από το προσκήνιο. Ελπίζουμε όταν θα έχετε λίγο να παυθεί να μπορέσετε να συνεχίσετε να συνεισφέρετε. Και σίγουρα τα μέλη της Επιτροπής μας θέλουμε να, θα ήθελα να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους για την διάθεση του χρόνου μας για τους τελευταίους ε, μήνες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. If, if you could return to your seat. Παρακαλώ να επιστρέψετε στις θέσεις σας. Λοιπόν, όσοι έφυγαν και όσοι αποχωρούν και αποχαιρέτησαν τον Ζαν Κλοντ μπορούν να επιστρέψουν. Ευχαριστώ. Τώρα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στην οδηγία Omnibus 2. Πρέπει να θυμηθώ και να υπενθυμίσω ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω έλλειψης χρόνου πρέπει να ακούσουμε, επειδή δεν μπορέσαμε να ακούσουμε, τη θέση, την τοποθέτησή της ε, ε, και ε, θα πρέπει εδώ αυτή η δυνατότητα να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Θα δώσω τον λόγο φυσικά στον εισηγητή πρώτα, τον κύριο Μπούκαρτ Μπάλτς. Παρακαλώ ησυχία γιατί δεν μπορούν να κραυγάζουν οι εισηγητές Παρακαλώ κύριε Μπάλτ, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σίγουρα θα μεριμνήσω και θα προσέξω ώστε ο εκπρόσωπος ε, της Επιτροπής σήμερα να μπορέσει να λάβει τον λόγο και να παρέμβει σήμερα. Και για μένα προσωπικά που είμαι εισηγητής είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για την έκθεσή μου, Πρόεδρε, 180 περίπου τροπολογίες κατατέθηκαν τα κέντρα βάρους και νομίζω συμφωνούμε ήδη προηγούμενα είχαν προαναγγελθεί ποια θα είναι. Αφενός βέβαια αφορά το πρίμα φερεγγιότητας ε, όσον αφορά τους κινδύνους. Δεύτερον, το θέμα προσωρινής αντιστήχησης με τρίτα κράτη. Και φυσικά η ε, προθεσμία και οι όροι για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Τώρα για μία ακόμα φορά συζητούμε την ε, συνήφανση αυτών των διατάξεων. Όπως γραπτός ήδη έγινε και εγώ ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσωρινή τελική διατύπωση αυτών των διατάξεων όσο το δυνατόν νωρίτερα να την υποβάλει το χρονοδιάγραμμα για τις αρχές Οκτωβρίου έχει ήδη περάσει, έχει ήδη καταστεί ένα εδαφικό, είμαστε στις 11 Οκτωβρίου. Πιστεύω όμως για τις εκτελεστικές διατάξεις 400 σελίδων θα πρέπει να, εξεταστεί επαρκώς από πλευράς μας. Προτού στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή καθορίσουμε τις θέσεις μας. Αν οι συνάδελφοι έχουν παρόμοια αξιολόγηση ή τελείω διαφορετική, με ενδιαφέρει το feedback, να ακούσω τις απόψεις τους. Σύντομα, δύο λόγια για την οδηγία πλαίσιο και τις εκτελεστικές διατάξεις. Όπως ε, στο σχέδιο έκθεσης ε, εκθέτω την άποψη το δυνατόν περισσότερα πεδία να καλυφθούν, ιδιαίτερα όλα τα πολιτικά σημαντικά θέματα στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου και να κατοχυρωθούν έτσι. Άλλοι συνάδελφοι πρότειναν μια άλλη πορεία. Δική μας δουλειά είναι τώρα να αποφασίσουμε αν την συναπόφαση ως εξουσία θα την ενδυναμώσουμε και στους εμπλεκόμενους στην αγορά δώσουμε ταχύτερα μια νομική ασφάλεια όπως την χρειάζονται. Η δική μου πορεία και προσέγγιση για την ταξινόμηση των εκτελεστικών διατάξεων σε κατεντολήν πράξης και τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης και προδιαγραφών δεν είναι κάτι που υπέστη επικρίση ως αυτός σκοπός. Γι' αυτό παρακαλώ δώστε μου τις απόψεις σας σήμερα, αν παρερμήνευσα κάποια πράγματα η προσέγγιση μου ανταποκρίνεται ακριβώς σε εκείνα τα οποία ήδη στο Omnibus 1 με εισηγητή τον Σάντσες Πρεσέντο είχαμε αποφασίσει και βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με αυτά που το Κοινοβούλιο υπό μια ισχυρή δομή ευρωπαϊκής εποπτείας είχε προτείνει δεν παραμέλησα τις φωνές και τις παρεμβάσεις που θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμα όριμη για τέτοιου είδους φιλόδοξα εγχειρήματα. Με ενδιαφέρον αλλά και με ερωτηματικά έχω αντιμετωπίσει το θέμα του, α, της ε, ρήτρας ε, εκπνοής. Εδώ θα πρέπει να συζητηθούν κάποια πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος και εδώ θα ήμουν ευγνώμων αν οι συνάδελφοί μας ε, γνωστοποιούσαν τις απόψεις τους. Και τώρα για το πρίμ φερεγγιότητας η εξέβρεση συμβαστική λύσης σίγουρα θα είναι πρόκληση για μας όλους. Κάποιε ε, τροπολογίες αντικαθιστούν το πριμ φερεγγιότητας ή ρευστότητα ε, με ένα πριμ αντικυκλική μορφή ε, που θα αντανακλάται. Άλλες τροπολογίες συμπληρώνουν το matching ε, πριμ. Άλλοι παραμένουν στο πριμ ε, ρευστότητα, αλλά θέλουν λιγότερο περιοριστικό να είναι το πλαίσιο εφαρμογή. Και άλλοι προτείνουν μια τελείω άλλη, διαφορετική προσέγγιση όπως της ε, αντικυκλικής αντιμετώπισης. Για την προσωρινή αντιστήχηση είμαι ανοιχτό να συζητήσουμε για τη λίστα κριτηρίων. Πώς προϋπόθεση για την εφαρμογή των προσωρινών αυτών αντιστοιχήσεων θα ισχύει μια ευρύτερη συνένεση φαίνεται να υπάρχει για την προσέγγιση της ε, μονοετούς ε, phasing in διάρκειας, όπως είχα και προτείνει. Και οι μεταβατικές διατάξεις ε, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν επιβεβαιωθεί ως προσδοκίες στις μεταβατικές διατάξεις και προτάσεις για το, τα κεφάλαια, για τις ομόλογα κτλ ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις ε, συμβιβαστικά και κάποιες άλλες παρατηρήσεις τώρα. Στοχεύω σε όλους τους συναδέλφους ε, που έχουν καταθέσει τροπολογίες γραπτός ε, να υποβάλω προτάσεις συμβιβαστικών τροπολογιών και είμαι πρόθυμος για προσωπικές συναντήσεις και συζητήσεις, ιδιαίτερα φυσικά με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ θερμά πρόεδρε. Καταρχά, θα περάσουμε στου σκιώδει ηγητέ. Δίνω καταρχά το λόγο στον Πίτερ Σκίνερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χάρη στις, ε, στα σκελισμένου ε, υπάρχει καλή ε, δουλειά των εισηγητών. Το τονίζω ιδιαίτερα, είναι εξαιρετικά καλό. Κατανοεί τα θέματα και κατανοεί επίσης και το κατεπήγον της υπόθεσης, αλλά επίσης κατανοεί και την ανάγκη να υπάρχει σωστή συζήτηση των θεμάτων. Η σχέση μεταξύ της εφαρμογής ε, μέτρων και της οδηγίας Omnibus 2 είναι ε, πάρα πολύ στενή, αλλά και η εφαρμογή των, με την εφαρμογή των μέτρων ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Omnibus 2 και την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων και πρέπει να δούμε πώς θα γεφυρώσουμε είναι σημαντικό να δούμε ότι με υπόβαθρο την οδηγία Solvency 2, που υπερψηφίστηκε μετά από πάρα πολλές αντιμαχίες, νομίζω ότι κάπου τέθησαν ε, αμετακίνητες κάποιες βασικές αρχές. Επί σειρά ετών ευελπιστούσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαβούλευσης να καταλήξουν, αν θέλετε, στο σκελετό στο ξύλο σκελετό του όλου οίκου, τον οποίο προσπαθούμε να κατασκευάσουμε για να προχωρήσουμε σε όλε τι συζητήσει και να πούμε ότι η πω πρέπει να περάσει συγκεκριμένο νόμο στο σύνολο των 27 χωρών τη Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμέναμε ήδη όμω επί μακρόν. Ο Μπέρκετ έχει δίκιο. Πλέον υπάρχει ανυπομονησία, ανυπομονησία από πλευρέ μα. Θέλουμε να δούμε πλέον αν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά ε, όταν βλέποντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται με συγκεκριμένα εφαρμοστικά μέτρα με μέχρι το τέλο του μήνα. Έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να αντιπαραβάλουμε τις προτάσεις της Omnibus 2 με τις συζητήσεις επί των τροπολογιών που είχαμε στο παρελθόν. Οφείλω να πω λοιπόν ότι αυτό καταρχάς. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι σε σχέση με αυτά έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες που εάν ε, υλοποιηθούν όλα αυτά μπορεί να οδηγήσει στις προσαρμογές που θέλουμε σε σχέση με την δουλειά γεφύρωσης που χρειαζόμαστε μεταξύ των μέτρων εφαρμογής και της ε, Omnibus 2 φαίνεται, αν θέλετε, να είναι συνολικά η δουλειά μας, αλλά υπάρχουν κανένα δύο άτομα στην αίθουσα που το κατάλληλο απολύτως. Έχω βάλει και μια συνοπτική ρήτρα που επιτρέπει ενδεχομένως να φερθεί η εργασία την οποία κάνει η Επιτροπή και να τη βάλει στα μέτρα εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα θα αναφέρονται και απαραίτητες νομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε για να αντικατοπτρίζονται οι σωστές αλλαγές στην Omnibus 2 σε σχέση με τις συνθήκες Λισαβόνας. Δεν θέλω να αναπτύξω συγκεκριμένα τις τροπολογίες μου, απλώς θέλω να σας πω ότι αυτό μας δίνει κάποιο βαθμό αξιοπιστίας στην, ε, απέναντι στην ε, κοινή γνώμη, πέρα από το Κοινοβουλίο και επίσης βάζει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματικά στο, σε προσοχή για να καταλάβουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, βλέπει πάρα πολύ σημαντικά το έργο και το ρόλο του, αλλά θέλουμε βέβαια να επιταχύνουμε βάζοντας, αν θέλετε, δίπλα-δίπλα αυτά τα δύο θεσμικά όργανα, αντί να περιμένουμε να έρθει το καθένα με τη σειρά του αντιμετώπιση του θέματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιλβί, από του Λευθέρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω μετά από όσα είπε ο Πίτερ. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να δουλεύουμε μαζί, το ξέρετε. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την δουλειά και για όλα αυτά που θα κάνουμε μαζί στο μέλλον και ευχαριστώ εκ των προτέρων. Είμαι μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει προτάσει σε ό,τι αφορά το πριν ρευστότητα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε το μάθημα από την κρίση την οποία βιώνουμε. Δεν διατείνομαι ότι έχω την λύση, κάθε άλλο. Είμαι ανοιχτή συζήτηση με όλου του συναδέλφου. Λέω απλώ ότι δεν θα πρέπει να, να βλέπουμε τι περιόδου αυτή τη κρίση που βιώνουμε, που είναι εξαιρετικά δύσκολου, ε, να μην τι παρακάπτουμε. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια σωστή λύση. Ταυτόχρονα το άλλο ζήτημα το οποίο με προβληματίζει είναι το πέρασμα κάποιων χαρτοφυλακίων από το ένα στο άλλο. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη μετάβαση, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να δούμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείε μπορούν να εξαφανίζονται από την αγορά, αν θέλετε, ενώ ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μακρόπνοους επενδυτές, περισσότερο από ποτέ. Χωρί να επισέρχομαι λοιπόν στα τεχνικά ζητήματα, υπάρχουν κανένα δύο ζητήματα πάνω στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και να δούμε στη συνέχεια πώ θα τα αντιμετωπίσουμε από τεχνική υφή. Δεδομένου βέβαια ότι όντω πρόκειται για κείμενα τα οποία είναι εξαιρετικά τεχνική υφή, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δουλειά που έγινε προηγουμένω για την οδηγία Omnibus 1 και να δούμε στο πνεύμα αυτό τι προσπαθούμε να κάνουμε για να υπάρχει συνοχή σε ό,τι αφορά του εμπλεκόμενου ε, ε, Εν πάση περιπτώσει, σα έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Το λέω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσλι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο για τη δουλειά του σε ένα πολύ δύσκολο και τεχνικό ζήτημα. Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα όλοι συμφωνούμε πως για τη φερεγγιότητα 2 πρέπει να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν και δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά στο σχέδιο εφαρμοστικών μέτρων. Γι' αυτό υποστηρίζω την τροπολογία σας 299 για να αποφευθούν ακριβώ καθυστερήσεις. Δεύτερον, θα πρέπει ο κλάδος να έχει μακροπρόθεσμη βεβαιότητα όσον αφορά την ισοδυναμία με τρίτες χώρες. Ο ασφαλιστικός κλάδος δουλεύει μακροπρόθεσμα και πρέπει να τους δοθεί μια κάποια βεβαιότητα πέρα από τα πέντε χρόνια. Γι' αυτό έχω καταθέσει τροπολογίες που δίνουν εξουσία στην Κομισιόν να επεκτείνει την ε, περίοδο την προσωρινή μετά από ε, μια αξιολόγηση κατά πέντε ακόμα έτη. Επίσης, στο 172 και στο 227 τα άρθρα έχω καταθέσει τροπολογίες έτσι ώστε να μπορούν να υποφιληθούν από τα της ισοδυναμίας και ευρωπαϊκές εταιρείες και όχι μόνο εταιρείες τρίτων χωρών. Επίσης έχω ε, καταθέσει και τροπολογίες για το ποια θα πρέπει να είναι η έκπτωση και μία ε, στάνταρ φόρμουλα για ένα πριν το οποίο θα είναι βεβαίως ε, είτε κυκλικό είτε μη υπομορφή ρευστού πράγματα, που φαντάζομαι είναι συναρπαστικά για τους υπόλοιπου ε, συνάδελφους. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε, αρκεί να αποτελέσει μια πρακτική λύση. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Μπέρκαρτ και τους υπόλοιπους ε, ηγητές για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Σβέν. Πρώτα απ' όλα και από πλευρά μου θερμές ευχαριστίες για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Ήταν πραγματικά κάτι που μας ε, ικανοποιεί και ικανοποίησε και ελπίζω ότι όλα έτσι θα προχωρήσουν. Για κάποια βέβαια από τα ζητήματα δεν θα είναι τόσο απλό αυτό, δεδομένων των διαφορετικών θεμάτων να εξευρεθούν κάποιοι συμβιβασμοί. Εγώ πιστεύω ότι το σημείο που είναι ενδιαφέρον είναι πόσο μεγάλο θα είναι το ενδιαφέρον σε σχέση με κάποιες ειδικέ έκτακτες ρυθμίσεις σαν αποτέλεσμα κρίσης. Το πριμ ρευστότητα, το matching πριμ, το αντικυκλικό πριμ, η ιστορία αυτών των πριμ είναι πραγματικά επιφανής, εξοχότατη. Ξεκίνησε με την ασφαλιστική, ε, τις ασφαλιστικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαν πρόβλημα με το πριμ ρευστότητα. Μετά δεν υπήρξε μεγάλη ικανοποίηση. Μετά σημείωσε η Ισπανική ασφαλιστική βιομηχανία ότι είχε πρόβλημα. Και τελικά για να επιληθεί το κοινό πρόβλημα εξευρέθη ένα matching prim ως πριν. Δυστυχώς δεν υπήρξε και υποστήριξη άλλων κρατών μελών, διότι αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό και ειδικό. Όταν διαπίστωσαν οι Ιταλοί ότι είχαν και εκείνοι πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα, καταλήξαμε στο αντικυκλικό πριν, πολύ ωραία. Τώρα αυτό βρήκε μια ευρύτερη υποστήριξη γιατί κάποτε όλα τα συμφέροντα των τομέων καλύφθη, καλύφθηκαν και εξυπηρετήθηκαν. Και τώρα, κορονίδα του στέματος, θα χάσει η Ευρώπη το δικαίωμα να αξιολογεί και να κρίνει σε ποιο σημείο η κατάσταση αντιμετωπίζει ένταση και πίεση και όλα με κάποιο αυτόματο αυτοματισμό τρόπο θα επιληθούν. Πρέπει να πω εξαιρετική δουλειά έκαναν οι λομπιίστες, εξαιρετικά δούλεψαν πέρα από σύνορα κρατών μελών. Μπορώ να κατανοήσω βέβαια ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου οι τιμές τη αγορά δεν δείχνουν, δεν αντανακλούν την αλήθεια και γι' αυτό υπάρχουν και προβλήματα. Δείχνω κατανόηση γι' αυτό σίγουρα, όμως υποστηρίζω αυτό που ο Μπούρκαρτ Μπάλτσε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ήδη είπε, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην εξυπηρετούμε ειδικά ιδιωτελή συμφέροντα και να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να εξαλήφωνε, να μην λαμβάνονται υπόψη. Τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον είδα ότι υπάρχουν άλλες ειδικέ επιθυμίες και έκτακτα πράγματα, ιδιαίτερα να αναφερθούν τα συμφέροντα των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ε, ασφαλιστικών εταιριών ασθένειας που έχουν κάποιο πρόβλημα τώρα. Θα επιθυμούσα, ήθελα και θα το επιθυμούσα με κάθε σοβαρότητα να τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, να συνέρθουμε και συνολικά, σφαιρικά να αναλύσουμε ποια είναι τα προβλήματα αυτή τη κρίση. Αυτό δεν μπορεί με συσσόρευση ειδικών επιθυμιών να γίνει και ει βάρο των ασφαλιζόμενων. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο το οποίο αφορά την υπέρμετρη χρήση των πριμ και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τι γίνεται με την προστασία όσον αφορά αντικυκλικές ε, εξελίξεις ε, και για τέτοιου είδους ε, κυκλικές τρευλώσεις τι μπορεί να γίνει. Θα ήθελα να είμαστε ισορροπημένοι στη συζήτηση και έχω την εντύπωση ότι ακριβώς ο εισηγητής στο δικό του σχέδιο προσπαθεί να επιτύχει αυτή την εξισορρόπηση πραγμάτων θα έλπιζα, θα επιθυμούσα παρόλες τις τροπολογίες ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε η προσπάθεια να επιτευχθεί, να κατευθυνθούμε όλοι προς την κοινή αυτή κατεύθυνση προς όφελος των ασφαλισμένων. Υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Financial Times σήμερα για τη Γερμανία και εν ώψη αυτής της εξέλιξης και έλεγε ότι είναι προ όφελο όλων των εμπλεκόμενων, όχι όμω των ασφαλισμένων. Θα ήθελα στο Κοινοβούλιο πρώτα οι ασφαλισμένοι στα συμφέροντά του να ληφθούν υπόψη. Σε εξισορρόψη συμφερόντων όσον αφορά εκείνου που προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα. Αλλά αυτό πρέπει να έχει κάποια αρχή, τέλο και ισορροπία. Και βλέπω ότι αυτά έχουν απολεστεί εδώ. Και με ενδιαφέρον διαπίστωσα ότι δεν ισχύει για όλου αυτό. Υποστηρίζουμε τις τροπολογίες ρητά της Σιλβί Γκουλάρ 344, 45, 46 που προσπαθούν αυτά τα θέματα, δηλαδή να υπάρξει μια διακοπή όσον αφορά ε, των κεφαλαίων asset και υποχρεώσεων, liabilities. Και αυτό το οποίο ε, προτείνεται βρίσκει πλήρη υποστήριξή μας. Πέρα από όλα αυτά δεν θέλω τώρα να ξανανοίξω όλα τα θέματα στη συζήτηση, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε και θα έπρεπε στενά με τα θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις και συλλόγους προστασίας των καταναλωτών και την ασφαλιστική βιομηχανία να συζητήσουμε. Αλλιώς θα χάσουμε και την αρχή και το τέλος και τη μέση και την ισορροπία. Και θα ε, κάνουμε κάτι όπως και για τα hedge funds. Δηλαδή θα μας γύρουν κατηγορίες, θα μας κατηγορήσουν ότι δεν ελήφθη υπόψη ο σκιώδης τραπεζικός τομέας κτλ. Λοιπόν, με παράλληλη πορεία να κινηθούμε όσον αφορά και για την, ε, το έργο που κάνουμε για τις τράπεζες. Να συναγάγουμε τα συμπεράσματα από αυτή την κρίση. Είμαι σύμφωνος με αυτά που λέει η Σίλβη. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα εκεί. Ευχαριστώ. Mr. Porter... Κύριος εδώ. Θα μιλήσετε Ναι. Ο Μίγκελ Πόρτας για λόγους υγείας απουσιάζει. Μου έστειλε ένα σύντομο κείμενο στα αγγλικά το οποίο θα ήθελε να διαβάσω η αγορά των ασφαλειών έχει ειδικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από το ότι τα περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι υποχρεωτικά και σχετίζονται με βασικές αποφάσεις. Αυτό καθά ακόμη περισσότερο αναγκαίο το να υπάρξει μια αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και ολόκληρη της οικονομίας. τεθεί έμφαση στην ε, βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών είναι κάτι το οποίο δεν προσφέρει καμία διέξοδο. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να έχουμε πελάτες ασφαλιών με αρκετή πληροφόρηση και πείρα για να αναλύσουν παραδείγματος χάρη τη και τη σταθερότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συναλλάσσονται. Αυτό σημαίνει πως η οι αλλαγές στον ευρωπαϊκό εποπτικό ρόλο και η ανάλογη εποπτική προσπάθεια πρέπει να γίνεται στο επίπεδο της Ευρώπης. Το να μην γίνει αυτό θα δυσκολεύσει τις χώρες οι οποίες έχουν απαιτητικά καθιστώτα και θα τις αναγκάσει να απορριθμίσουν ενώ θα ωφελήσει τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούν σε Χώρε με λιγότερο αυστηρού κανόνε. Ένα από τα βασικά ζητήματα στη συζήτηση αυτή είναι οι πληροφορίε οι οποίε θα πρέπει να υποβάλουν οι εταιρείε εθνικέ εποπτικέ αρχέ. Θα είναι ένα βήμα προ τη λάθο κατεύθυνση να χαλαρώσουν οι υποχρεώσει των εταιριών όπω η υποχρέωση να υποβάλουν έναν πλήρη κατάλογο στοιχείων ενεργητικού σε τακτική βάση. Οι ευρωπαϊκές χώρες με τις καλύτερες ε, ρυθμιστικές ε, πρακτικές. Ε, αυτός ο κατάλογος πρέπει να υποβάλλεται κάθε τρεις μήνες. Αυτά τα οποία λέγονται περί είναι υπερβολικά καθώς πρόκειται για πληροφορία την οποία πρέπει να έχουν ούτως ή άλλως οι εταιρείες. καθώς ε, αυτές ε, οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τις εποπτικές αρχές για να γίνει ανάλυση κινδύνου, θεωρούμε πως το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να ε, ρυθμίσει σύμφωνα με το ίδιο σετ κριτηρίων της απαιτήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε. Ζαν Πολ Καταρχάς, κυρία Πρόεδρε, να συμμεριστώ και εγώ τα εγκόμια προς τον συνάδελφο και παρακαθήμενο. Ε, όντας και τόσο κοντά της θέλω να είμαι πάρα πολύ ευγενής μαζί του. Αλλά θέλω βέβαια και να χαιρετήσω ιδιαίτερα και να το συγχαρώ για την εργασία του και να υπενθυμίσω κάποια σημεία τα οποία είναι σημαντικά κατά μένα είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη καταρχάς την προστασία των ασφαλισμένων. Είναι εξίσου σημαντικό η ευρωπαϊκή, ο ευρωπαϊκός τομέας ασφαλίσεων να μην κυρωθεί. Ε, έχουμε την τάση να είμαστε εξαιρετικά αφελείς των τρόπων τον οποίο νομοθετούμε. Έχοντας λάβει διάφορα μέτρα εξαιρετικά δεσμευτικά, τελικά δεν τα εφαρμόζουμε. Και το υπογράμμισα προηγουμένως και στον κύριο Τρισέ κάποιες ε, παρατηρήσεις. Καταρχάς, η μετάβαση σε ό,τι αφορά την ε, ισοτιμία με τρίτα μέρη. Δεν θα πρέπει να ακυρώσουμε θυγατρικές ευρωπαϊκών εταιριών που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, ε, επιτρέποντας τους να εφαρμόζουν τους τοπικούς νόμους και κανόνες, οπότε μπορούν να βρουν σχετική ισοτιμία. Πρέπει να υπάρξει κατάλληλος χρόνος γι' αυτό. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την μεταφορά κάποιων ε, μετοχών. Ξέρετε, τα χρηματοστατικά ιδρύματα βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στα χρηματοοικονομικά του, σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο των ε, χρεογράφων του. Θα πρέπει να αποφευχθεί σε περίοδους κρίσης που διανύουμε όπω αυτοί οι εταιρείε αυτέ να οδηγηθούν, να διαφοροποιούνται στι αγορέ, να εκποιούν γρήγορα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν, το οποίο οδηγεί και σε μείωση των τιμών και δεν δίνεται δυνατότητα να λάβουν τις ε, κατάλληλες και σωστές αξίες τις οποίες έχουν ε, υποσχεθεί άμεσα ή έμεσα ασφαλισμένους. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ασφαλιζόμενους, πρέπει οι ασφαλιστές να είναι ισότιμοι με τα ιδρύματα τα οποία διέπονται από την εξειδικευμένη αυτή οδηγία και μέχρι ότου η οδηγία επικαιροποιηθεί και εξυγχρονιστεί, θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε τοπικές στρεμπλώσεις ανταγωνισμού. Τέλος, δεν θα εκπλαγείτε λέγοντάς σας ότι επιθυμώ οι Ευρωπαϊκές Ευρωπαϊκές Αρχές, η ΕΙΟΠΑ, να μην αποδυναμωθούν στον διαιτητικό τους ρόλο, ώστε να μην υπάρξει dumping καονιστικό και να υπάρχει ασυνέχεια και ασυνέπεια ε, μεταξύ των διαφόρων θεσμοθετών και υποπτικών αρχών στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αν και ο κανονισμός Omnibus 2 είναι εξαιρετικά τεχνικής φύσης, ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά πολιτικής ε, φύσης, γιατί ως κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια θέλαμε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πλαίσια που δίνουν σημαντικό ρόλο στους Ευρωπαίους επόπτες και είμαστε ευγνώμονες ε, στην εργασία που επιτέλεσε Book of στην έκθεση αυτή, συνεχίζοντας αυτή την προηγούμενη πορεία που έχει χαράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί και πάλι βέβαια θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ισχυροί και συνεπείς στην ε, προσέγγιση μας. Και χάρη στην ε, έκθεση την οποία συντάξατε, νομίζουμε ότι όντως κινείται σωστή κατεύθυνση. Πολύ ισχυρό ο ρόλος λοιπόν για τον ε, ΑΕΟΠΑ Πρέπει να δούμε βέβαια και τα πρακτικά ζητήματα, γιατί θέλουμε ταχύτητα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και να τηρήσουμε τις αρχές μας. Είμαστε όμως σε πολύ καλά χέρια, στα καλά και στιβαρά χέρια του Μπούρκαρτ, για να βρει τη σωστή ισορροπία. Τώρα, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Υποπτικού Οργάνου της ΑΕΟΠΑ μπορεί να το συζητήσουμε σε ό,τι αφορά το κυκλικό premium σε εποχές κρίσης των χρηματοοικονομικών αγορών. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα γιατί κατα... Ε, υποβάλλατε την τροπολογία 77 όπου περιλαμβάνεται και τη διάταξη ότι ο εθνικός νομοθέτης θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα premium ρευστότητα ε, από τους ε, ασφαλιστές. Και γιατί να, μην το, να το επιτρέψει αυτό και να το αποφασίσει ο ΙΟΠΑ. Γιατί το αφήνεται στη διακριτική αρχή στη διακρίτηση των ε, εθνικών αρχών. Δεν θα πρέπει να εισάγουμε κάποια προδιαγραφέ σε αυτό, το θέμα. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί σωστή λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους, ε, ε, την ασφάλιση υγείας, θέλω να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά όταν πρόκειται περί εξαιρέσεων, είναι εύκολο να πούμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των, των ασφαλιστών των ασφολιστών και ότι ασκούν πίεση γι' αυτό. Έχουμε όμως και τα συμφέροντα των ασφαλιζομένων. Για παράδειγμα, στις κάτω χώρες έχουμε πολύ ισχυρούς ε, κυβερνητικούς κανονισμούς σε ό,τι αφορά το, τους κινδύνους και τα συστήματα εξισορρόπησης που υπάρχουν και είναι από τη σκοπιά του συμφέροντος των ε, ασφαλιζομένων που αναγνωρίζεται και στο κοινοτικό σύστημα. Γιατί διαφορετικά θα τα με πολύ πιο υψηλά ασφάλιστρα. Γιατί τότε θα πρέπει να διπλοπληρώσουν για την ανάληψη, για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου. Και αυτό αναγνωρίζεται και από τον ε, εισηγητή. Πρέπει να δούμε δηλαδή και την πλευρά του ασφαλιζόμενου σε αυτό το πεδίο αλλά βέβαια είμαι πρόσφορη και ανοιχτή σε σχετική συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ισοτιμία τρίτης χώρας, συμφωνώ με αυτό που είπε ο εισηγητής Κιουμπούκου, πρέπει, το είδαμε και από το Νομισματικό Ταμείο, πρέπει να έχουμε σαφείς αρχές. Και εγώ προτιμώ την, ε, μια, προτιμώ μια σύντομη μεταβατική περίοδο, αλλά χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να δουλέψει και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία αλλά νομίζω ότι και σε αυτό ο Μπούρκαρτ ε, είναι στον, σε σωστή πορεία και μπορούμε να το εξειδικεύσουμε αυτό και να βρούμε τις σωστές ε, λύσεις. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι το καλύτερο στην, ε, σε ό,τι αφορά την τύχη των συμβαστικών τροπολογιών και ελπίζω να υποστηριχθούν από μεγάλη πλειοψηφία. Είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε την γραμμή σας σε ό,τι αφορά το ρόλο των εποπτικών αρχών γιατί διαφορετικά μπορούμε να βρεθούμε πάλι σε διαπάλλη με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αν τον ανέχει το λόγο. Ο κύριος Σάντσες Πεσέδο παρακαλώ. Και εγώ θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου για το ότι ο κύριος Μπάρς εισηγητής θα μπορέσει να βρει επαρκή επίλυση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το θεμελιώδες ζήτημα είναι η σπουδαιότητα των ε, θεμάτων. Αν όλα αυτά είναι επαρκώς ε, ικανά ή αν θα πρέπει αν υπάρχει εποπτεία, επόπτης ο οποίος ε, θα δρά. Είναι θέματα σπουδαιότατα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θεωρούμε ότι είναι σπουδαία και πρέπει έτσι να αντιμετωπιστούν. Συζητάμε αν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστούν ή όχι. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, επειδή μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Και γι' αυτό μπορεί να υπάρξει, αν δεν γίνει κάτι σωστό, μια μεγάλη διατάραξη στη μεταβατική περίοδο. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία στη λειτουργία του συστήματο όπω είναι ευκταίο. Και δεύτερον, για λόγου αποτελεσματικότητα. Μπορούμε να συζητήσουμε αν θα είναι αντικείμενο αυτών των θεμάτων ή κάποιες διατάξεις που θα εξεταστούν για να μην υπάρχει κάποιος ξεχωριστός χαρακτήρας, έκτακτος χαρακτήρας. Το θέμα είναι σπουδαίο, σημαντικό και για τους εξής λόγους. Για τις κυκλικές περιπτώσεις και κυκλικές εξελίξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ιδιομορφία τους. Θα πρέπει στην εποπτεία να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τη μεγάλη μεταβλητότητα η μεγάλη μεταβλητότητα, ευμεταβλητότητα μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές σε πολύ σύντομες χρονικές περιόδους. Γι' αυτό πρέπει να αποφύγουμε οι εταιρείε να βρεθούν σε τεράστια τέτοια πίεση από τον ευμετάβλητο χαρακτήρα των εξελίξεων. Αυτό το στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον επόπτη, από την εποπτεία. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή που είναι πολύ σημαντική πιστεύω εγώ και προέρχεται όσον αφορά τις υποθήκες, τα ενυπόθηκα δάνεια. Είναι στοιχείο κλειδί για τη μέγιστη ισορροπία όταν τα ενεργά, τα κεφάλαια και οι υποχρεώσεις πρέπει τα ίσεις ίδιες προθεσμίες ε, να, έχουν, να μπορούν να αντιστοιχούν η μία στην άλλη. Μακροπρόθεσμα ή ε, ε, μεσοπρόθεσμα. Όταν έχουμε μακροπρόθεσμη κάλυψη, όταν έχουμε την ανάγκη να υπάρξει άμεση χρηματοοικοδεπτική κάλυψη, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα. Όταν έχουμε μεγαλύτερες ε, απαιτήσει ε, τις οποίες εισάγουμε υπάρχουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, μεγαλύτερο βάρος το οποίο υφίστανται οι εταιρείε. Γι' αυτό είναι δύο κριτήρια τα οποία είναι πάρα πολύ σχετικά και σημαντικά και όχι μόνο για τις ασφαλίσεις αλλά και για τη συνολική απάντηση που θα πρέπει να βρούμε και να δώσουμε συνολικά στην μεταρρύθμιση την ε, χρηματοοικονομική, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Ευχαριστώ. Η Ελίζα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Μπάλση για αυτό το περίπλοκο σύνθετο και θα έλεγα κείμενο που καλύπτει πολλές πτυχές ε, περιεκτικά. Οι δύο μου ερωτήσεις στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση όπως έγινε από την κυρία Κορίν ε, Βόρτμαν Κόλπιο πριν τη συνάδελφο. Λέει ότι για πρώτη φορά εργαζόμαστε με τον ΑΕΟΠΑ και το Κοινοβούλιο είχε δραστηριοποιηθεί ενεργά στο να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ύπαρξη και λειτουργία αυτού του νέου θεσμικού οργάνου αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής. Λοιπόν, όσον αφορά συγκεκριμένα τώρα την τροπολογία σας υπαριθμό 53 για το άρθρο 35, το εδάφιο 35, φαίνεται ότι η αρχική διατύπωση όσον αφορά το 35 είχε ως εξής για το άρθρο 35 λέει ότι προτείνεται οι επόπτες να έχουν τις εξουσίες να καθορίσουν την φύση, εύρος και μορφή της ε, έκθεσης ε, εποπτείας σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες περιόδους. Είναι μια ευρεία προσέγγιση που θα λέγα ότι βαίνει καλώς. Στη συνέχεια υστερότερα προσθέτεται με το άρθρο 53 κάτι άλλο. Τι λέτε, λέτε ότι η έκθεση ή μάλλον για περιόδους μικρότερες ε, των 12 μηνών οι τακτές ε, εκθέσεις εποπτείας περιορίζονται σε σχέση με το εύρος των πληροφοριών, σε σχέση με την περίοδο ενός έτους. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε όμως πραγματικά τις επιδόσεις ε, ενός οργάνου και αν δεν υπάρχει υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος με την τριμηνιαία ή τετραμηνιαία έκθεση, το να περιορίζονται οι πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροφορήσετε μόνο αν εκδηλώνεται, ξεσπάει μια έκδηλη κρίση, ε, τότε η ποιότητα της ε, εποπτικής ε, εργασίας, του εποπτικού έργου περιορίζεται. Διότι δεν γνωρίζετε ακριβώς ποιες είναι οι επιδόσεις ε, ενός τέτοιου οργάνου συνολικά. Αυτή η περιστολή, η περιοριστική θα έλεγα ρύθμιση, ίσως μπορεί να είναι θα μπορούσε δυνητικά να ήταν ένας περιορισμός για την ποιότητα, στην κατανόηση των εξελίξεων. Είσαστε λοιπόν υπέρ του να μην διατυπωθεί έτσι και να αναμείνετε για να δούμε πρώτα την λειτουργία του εποπτικού μηχανισμού προτού επισέλθουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Θα συμφωνούσατε να μην υπάρχουν τέτοιοι αυστηροί περιορισμοί προτού δούμε τι γίνεται στην πράξη. Και δεύτερον, όσον αφορά την τροπολογία σας 54, εδώ το εξής. Ζητείτε εσείς σαφώς ε, λέτε να απαγορευτεί ε, η απαρίθμηση σε ένα κατάλογο των κεφαλαίων ή των αποθεματικών ε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης όμως αυτό είναι Ζωτική σημασίας για να κατανοήσει κανείς τι συμβαίνει και ποια είναι τα αίτια ενός προβλήματος που ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτός ο περιορισμός πάλι, τα κράτη-μέλη, και αναφέρομαι ως παράθεμα στην τροπολογία σας, δεν θα πρέπει να ζητούνται από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες ε, να υποβάλουν στις εποπτικές αρχές ε, ένα πλήρη κατάλογο αποθεματικών ή κεφαλαίων απαριθμώντας ένα προς ένα τα πάντα, κάτι τέτοιο νομίζω τροχοπεδί την ευρεία πλήρη πληροφόρηση που πρέπει να έχουν οι εποπτικές αρχές για να κατανοήσουν τι τεκταίνεται. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων, μετά από την ε, ε, διαβούλευση για το πώς ε, αισθάνονται οι αρχές, η εποπτική αρχή, αν αυτό κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι περιορισμοί αυτοί που περιορίζουν στο έργο. Το έργο και αυτό είναι κάτι καινούριο, το οποίο όλοι σε αυτό το κοινοβούλιο υποστηρίξαμε να υπάρξει αυτή η ενεργοποίηση. Αυτό θα ήταν λοιπόν υπονόμευση της σωστής λειτουργίας της εποπτικής αρχής και έτσι δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε τον, την ανάγκη για τέτοιου είδους ε, περιορισμούς. Πέρα όμως από όλα αυτά, θα έλεγα ότι γενικά η έκθεση είναι ένα ε, αφορά ένα πολύ τεχνικό θέμα, είναι πολύ σωστή και ε, περιεκτική και Απλά θα ζητούσα αυτά τα δύο θέματα να λάβετε υπόψη, να τα εξετάσετε. Ιδιαίτερα θα πρότεινα να ακούσουμε την ΑΕΟΠΑ για να ακούσουμε και να αναδούμε αν αυτό θεωρείται ως περιοριστικός όρος και ως σοβαρός περιορισμός στην δράση, δραστηριοποίησή τους ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποιες αρνητικές διεργασίες στην ε, εκτέλεση του έργου της αρχής αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο. Το εγώ, λέει η πρόεδρο. Αλλά εντάξει κάποιο άλλο. Προφανώ θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινώ εγώ καταρχά. Συμφωνώ με όσα είπε η Λίσσα. Αισθάνομαι ότι το θέμα της επο... η εποπτική αρχή θα πρέπει να έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που θεωρεί ότι είναι εκεί η σωστή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα θέτουν ερωτήματα επί παντός επιστητού πάντοτε αλλά πάντως θα ήταν λάθος να περιορίζονται, να περιορίζεται η οπτική αρχή αν αισθάνονται χρειάζεται κάποια πληροφόρηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ΕΟΠΑ θα έχει κάποιο ρόλο στο να είναι θεματοφύλακας ακριβώς αυτού του, αν θέλετε, του λογικού ή μη λογικού, αν υπάρχουν κάποιες υποδείξεις, κάποιες προτάσεις ε, εάν κάποια όρια έχουν υπερπηδηθεί ή αν υπάρχει κάποια υπερβολική επιβάρυνση, αν έχουν γίνει τα πράγματα κατά λάθασμένο τρόπο ή που, κατά τρόπο που ενδεχομένως θα μπορούσε να ε, παρέμβει και να στατώσει την ενιαία αγορά. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποια εποπτική αρχή να ζητά σχετική προφόρηση σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείε και να παραμποδίζει για κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα εφαρμογής ε, κανονισμών και χώρηση του θέματος. Το συζήτησα τελευταία φορά. Προφανώς χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, ε, ροπή, αν θέλετε, που έχει πάρει το θέμα. Το συζητήσαμε και άτυπα, αλλά και το θίξαμε, το στην Επιτροπή, όταν ήταν εδώ ο πρόεδρος του ΑΕΟΠΑ. Νομίζω ότι λειτουργεί αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο υποπτικός αυτός μηχανισμός ε, δεν είναι έτοιμος ή υποβιβάζεται, αλλά είναι θέμα, αν θέλετε, ε, αυτή τη στιγμή ε, ε πιο εύρυθμης λειτουργίας. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποιο προσχέδιο κανονισμού ταυτόχρονα και έχω στείλει σχετική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσω να μας δοθεί το προσχέδιο αυτό το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αν ξέρουμε λεπτομερέστερα πού εστιάζουμε, θα λειτουργήσουν και καλύτερα. Ο πεπτικός ε, οργανισμός αυτός δεν μπορεί να ξεκινήσει και να ασκήσει τις εξουσίες του μέχρι ότου πραγματικά ε, εφαρμοστεί η Solvency 2. Και είναι κάτι κατεπήγον αυτό. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το ιστορικό της υπόθεσης, όπως το χαρακτήρισε ο ε, Σβέν. Όταν εκπονούσαμε τα θέματα Solvency 2, είχαμε αυτό το πρόβλημα με τα χρεόγραφα και τις ε, ενδεχόμενες απόσεις από την αγορά ή και όλων των παρεπόμενων κυκλικών επιπτώσεων που θα είχε κάτι τέτοιο. Και είχαμε τότε εκφράσει πάρα πολλές ανησυχίες ως προς το τι θα συνεπαγόταν αυτό, ε, αν υπήρχε πια πιο μόνιμη απόσυρση ε, επενδύσεων ε, σε αξιόγραφα είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό μάλιστα για τη Γαλλία, η οποία ε, εξέφρασε την ανάγκη ύπαρξης κάποιου είδους μαξιλαριού, αν θέλετε, ώστε οι ενδεχόμενες επενδύσεις σε αξιόγραφα και η απόσυρση να μην αντικατοπτρίζεται άμεσα στο κεφάλαιο, στην κεφαλοχική επάρκεια χρηματοσυντητικών ιδρυμάτων δεν είχαμε σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Γιατί λίγο πολύ ξέραμε ότι έπαιρνε να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε με την Solvency 2 και ξέραμε ότι ήταν πράγματα μη περατωμένα και άλλοι παράγοντε οι οποίοι δεν είχαν πλήρω κατανοηθεί στο, περίοδο, στο πεδίο αυτό και θα έπαιρνε να το ξανασυζητήσουμε και σε ό,τι αφορά το μαξιλάρι αυτό των κυκλικών φαινομένων ή κατά πόσο το ζητήματα του θετικού και παθητικού των ασφαλιστικών οργανισμών, πώς τα ήταν. Για να δούμε λοιπόν πώς αυτά μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα πρόθυμο εταίρο, η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να μεταβιβάζονται ταυτόχρονα και από κοινού, γιατί είναι αλληλένδετα. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε είναι οι ασφαλιστικές εταιρείε να, κάνουν αυτή τη μεταβίβαση και να μεταβιβάζουν αυτό το ε, θετικό και παθετικό σε ένα κάποιο είδους ε, ε, χρηματοδοτικό εργαλείο ή σε κάποιο φορέα ή ειδικού σκοπού που δεν θα ήταν όμως άμεσα υπόλογο. Οπότε οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, οι δικαιούχοι αν θέλετε να πλήττονται από κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε όλη αυτή τη νοητική διαδικασία μεταξύ των κυκλικών ε, αυτών, των κυκλικών ε, ε, μαξιλαριών, των μαξιλαριών σε ό,τι αφορά τις κινητές αξίες και τα ασφαλιστρά ρευστότητας. Το ειδικό μου ενδιαφέρον, αν θέλετε, το προσωπικό, είναι ακριβώς, το προσωπικό μου ενδιαφέρον αφορά στους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους. Αυτούς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Ο Πίτερ ε, ανέφερε αυτούς τους ε, παράγοντες ε, συσχετισμού, γιατί παραπονιόμουν συνεχώς κατά τη διάρκεια του Solvency 2, γιατί δεν κατανοήσαμε ακριβώς πώς ε, κάποια ιδιαίτερα μακρόπρόθεσμα γεγονότα και γενικές καταστροφές συνδέονται. Αντί λοιπόν να έχουμε κάποια πράγματα παγιωμένα στο παράρτημα, κάποια τα ε, αναθέσαμε, αν θέλετε, και τα αναβάλαμε για περαιτέρω σκέψη. Κάτι άλλο που δεν πραγματευτήκαμε πλήρως είναι το πώς αναγνωρίζουμε την εξειδίκευση. Αναγνωρίζουμε ότι η διαφοροποίηση είναι κάτι καλό για τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά το ίδιο είναι και η εξειδίκευση και η καλύτερη και πολύ στενή γνώση κάποιου παιδιού περιορίζει το ρίσκο ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συσχετίζεται πάρα πολύ ισχυρά. Το σώθεση 2 λοιπόν όντως ε, λέει ότι κάτι τέτοιο πρέπει να αναγνωρίζεται. Δεν ε, έθελο τυφλό σε σχέση με κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν, λέγοντας ότι όντως έχουμε κάποια ειδικά συμφέροντα εδώ. Δεν λέω ότι συμφωνώ με όσα έχουν προταχθεί, αλλά έχουν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώσο θα επιλύουμε το πρόβλημα της ε, αγοράς κινητών αξιών, θα πρέπει να έρθουμε στα θεμελιώδη. Ποια ήταν η βασική πρόθεση στο πρώτο κείμενο Solvency 1 και Solvency 2 στη συνέχεια. Και για να είμαστε ρεαλιστές, αντικατοπτρίζοντας ακριβώς το ποια ήταν η πραγματικότητα στην αγορά, ποια ήταν η πραγματικότητα των ε, κινδύνων και των παθητικού και των υποχρεώσεων που αντιμετωπίζαμε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως στις τράπεζες, όπου έχουμε ε, ενεργητικό απέναντι στο οποίο τις αθμίζεις με διάφορα δάνεια ότι έχεις. Το γεγονός με τις υποχρεώσεις στις ασφαλιστικές ε, εταιρείε που δεν ξέρεις πότε θα καταπέσουν, ε, είναι πολύ πιο σημαντικές και απαιτούν πολύ μεγαλύτερη πρόληψη κεφαλοχική επάρκεια από τις τράπεζες. Και εάν είναι αληθές αυτό, είμαστε ακόμα στην καμπύλη μάθησης. Και θα ήταν πολύ λάθος να κλείσουμε την πόρτα, όπου πιστέψτε με όποιοι ακούτε, κάπου στη χώρα σας, κάποια ασφαλιστική εταιρεία ξαφνικά θα ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει κάποια υποχρεώσεις σας, υποχρεώσει σε κάποιον ε, πελάτη της, σε κάποιον δηλαδή ψηφοφόρο μας, γιατί κάποιες πόρτες έχουν κλείσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε και το θέμα της ευελιξίας χωρίς βεβαίως να υποσκάπτουμε οτιδήποτε ήταν η αρχική πρόθεση του στη δύο σχέση με τη σταθερότητα. Πολλά θα μπορούσα να πω ακόμα, αλλά λίγο πολύ ότι είπα ανακεφαλαιώνει τα όσα συζητήθηκαν. Εξτρέφομαι λοιπόν τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάρολ, νομίζω δώσαμε αρκετά που ίσως θα ήθελες να σχολιάσεις και στη συνέχεια θα ξαναδώσουμε το λόγο βέβαια στον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω ευχαριστώντα τον εισηγητή για την εκθεσή του. Δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω μέχρι τώρα και θέλω να το κάνω εξ ονόματο Κομισιόν. Να ευχαριστήσω και τα μέλη τη Επιτροπή σα για τι προτάσει ε, που έκαναν, που προσπαθούν να αναπτύξουν νομοθεσία. Σωστή και βεβαίω αυτό είναι ο στόχο τη διαδικασία τις ε, οδηγίες για τη φιωρεγγιότητα 2 και συμφωνώ βεβαίως πως τη χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε ένα σύστημα που είναι σωστό για την προστασία των ασφαλισμένων, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος νομοθεσίας. Κύριε Πρόεδρε, ζητήσατε κι εσείς και ο Πίτερ Σκίνερ από την Κομισιόν ε, τα εφαρμοστικά μέτρα ε, τα φέρουμε στην επιτροπή σας και, και ο κύριος Μπάλτσερ επίσης. Μπορώ λοιπόν να σας πω πως θα τα έχουμε αυτά μέχρι το τέλος του μηνός, μέχρι το τέλος του μηνός γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη φάση της διαβούλευσης και πρέπει να τονίσουμε πως μας απασχολεί αυτό το θέμα εδώ και δύο χρόνια μαζί με την ΙΟΠΑ που μετά έγινε ΣΕΟΠΣ και αποτελεί τη βάση βεβαίως των σκέψεών μας και με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η διαβούλευση γιατί αποφασίσαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά για να αντιληφθούμε πλήρως ποια είναι τα ζητήματα και το εάν μπορούμε να βρούμε μια σωστή λύση. Μέχρι το τέλος του μήνα, κυρία Πρόεδρε, η Κομισιόν θα σας δώσει το κείμενο πρόχειρο, όπως είναι γύρω στις 400 σελίδες. Όσον αφορά τώρα τη διάκριση μεταξύ πράξεων ε, κατεξιοδότηση και τεχνικών προδιαγραφών. Πρέπει να τονίσουμε πρώτα απ' όλα πως η φερεγγιότητα 2 δεν μπορεί να συγκριθεί με την οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων γιατί η ε, οδηγία αυτή ε, έχει ισχυριστεί ακριβώ έτσι για να υπάρχει ένα επίπεδο 2 και ένα επίπεδο 3. Τώρα η πράξη κατεξιοδότηση που είχε προβλέψει η Κομισιόν θα πρέπει να ξέρετε πώς ε, ανήκουν στο πεδίο των τεχνικών προδιαγραφών, κάτι το οποίο δεν υπήρχε όταν σχεδιάζαμε τη φερεγγιότητα δύο, αλλά η Κομισιόν βεβαίως ευχαρίστως μαζί σας να σκεφτεί το πώς θα λύσουμε αυτό το ζήτημα. Νομίζω πως μια ρήτρα σταδιακής εισαγωγή μπορεί να αποτελέσει μια λύση. Να τονίσω επίσης πως με βάση τον κανονισμό για την ΕΖΑ δεν θα πρέπει οι τεχνικέ προδιαγραφέ να αποτελούν μια επιλογή πολιτική Είναι ακριβώ τεχνικέ προδιαγραφέ και άρα θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Η Κομισιόν είναι στη διάθεσή σα για να σα βοηθήσει αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο τη ΕΟΠΑ, η οποία βεβαίω παίζει σημαντικό ρόλο. Αναφέρθηκε η ισοδυναμία επίση. Η ισοδυναμία με τρίτε χώρε και ειδικά τα μεταβατικά μέτρα. Μπορώ να σα πω, κύριε Πρόεδρε, πω υπάρχουν πολλέ χώρε στον κόσμο που ε, εξετάζουν την φερικαιότητα 2 ως μέσο για να βελτιώσουν το νομοθετικό τους ε, πλαίσιο στην ε, Διεθνή Ένωση Ασφαλιστικών Επιτροπών. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω πολλές από αυτές τις χώρες για τη φερικαιότητα 2 και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι πως εμείς έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος να σκεφτόμαστε πως όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει προχωρήσει όσο εμείς. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί από αυτές τις τρίτες χώρες. Σημαντικό είναι λοιπόν να υπάρχει μια βεβαιότητα για τον κλάδο, ο οποίος είναι παγκοσμιοποιημένος και να βοηθήσουμε και τις χώρες αυτές στο να περάσει το πλαίσιο αυτό της φεργαιότητας σε μια κατεύθυνση που θα βασίζεται περισσότερο στον, στην αξιολόγηση κινδύνου. Και το πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με ένα μεταβατικό καθεστώς 5 ετών ή καλύτερο. Όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν. Αναφέρατε το θέμα του πριμ ρευστότητα που τώρα λέγεται αντικυκλικό πριμ, το matching πριμ κτλ. Κύρια Πρόεδρε, και εμεί τα ίδια ακριβώ είχαμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη και του ενδιαφερομένου. Αυτό το οποίο αναγνωρίσαμε, κύριε Γκίγκολτ, μετά την οικονομική κρίση, που μάθαμε, γιατί συνεχώ μαθαίνουμε, αναγνωρίσαμε πως πρέπει να προσέξουμε, να μην δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει τεχνητές αναταράξεις και άρα θα διαταράξει το βασικό ρόλο της ασφάλειας, δηλαδή μακροπρόθεσμες εγγυήσεις. Και αυτό δεν βασίστηκε σε κάποιο λόμπι. Ήταν μέρος μιας συνολικής εικόνας. Κοιτάξαμε την πλευρά των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί και πώς θα μπορέσουμε να μην διαταράξουμε την εικόνα όταν τα σπέρα στην αγορά ανεβοκατεβαίνουν στο Άγιο Γιο. Οπότε θα πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείε να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν αυτές τις ε, μακροπρόθεσμες ασφάλειες σε ένα τόσο σε ένα περιβάλλον με τόσο μεγάλες αναταράξεις. Γι' αυτό κοιτάμε αυτό το πριν, το αντικυκλικό που θα μπορούσε να λύσει αυτό το ζήτημα και βέβαια εδώ πέρα το θέμα είναι ποιος είναι ο ρόλος της ΕΟΠΑ. Κάποιοι θέλουν ε, μια προσέγγιση με έναν τύπο με το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε γιατί βεβαίως ε, αν γίνει αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αιτία της επόμενης κρίσης και να τη βάλουμε σε ένα τύπο. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε ποια κριτήρια θα πρέπει να συνοδεύουν την παρέμβαση της ΕΟΠΑ. Όταν, ε, πότε πρέπει δηλαδή να παρέμβει η ΕΟΠΑ για να αναπτύξουμε έναν τύπο όταν έχουμε αυτές τις ακραίες συνθήκες στην αγορά. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση για τα μεταβατικά μέτρα και συμφωνώ με τον εισηγητή πως πρέπει να τα περιορίσουμε αυτά μόνο στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε μεταβατικές ε, περιόδους όπου να έχουν πάλι διαφορετικές επιλογές στα κράτη-μέλη. Αν έχουν επιλογές τα κράτη-μέλη για να αποφασίσουν πως για μια σειρά ετών μπορούν να κάνουν το χ ή ε, το δώσουμε αυτό στην Εθνική Εποπτική Αρχή, ε, εμεί θα ήμασταν κατά. Γιατί έτσι δεν θα έχουμε μόνο 27 καθεστώτα, αλλά νη συνένα. Γιατί είναι πολύ εφευρετικά τα κράτη-μέλη στο να εφευρέσκουν διάφορου μηχανισμού για την βελτίωση της κατάστασής τους όπως πιστεύουμε. Γι' αυτό συμφωνώ με όσους είπαν εάν έχουμε μια μεταβατική περίοδο να αποφασίσει η ΕΟΠΑ. Όπως ε, ακριβώς και συζητάμε την ε, ασφάλιση υγείας, το αναφέρατε κυρία Βόρτμαν Κόλ στην Ολλανδία. Είναι σημαντικό το σύστημα για την Ολλανδία, το γνωρίζουμε, γι' αυτό ακριβώς σχεδιάσαμε ένα σύστημα με το οποίο η ΕΟΠΑ θα αποφασίζει το εάν θα πρέπει να υπάρξει μια εξαίρεση για την Ολλανδία σε στενή συνεργασία με την Ολλανδική Εποπτική Αρχή. Τώρα, για μετοχικά κεφάλαια, πράγματι υποστηρίξαμε μια μεταβατική περίοδο γιατί πράγματι βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο των αναταραχών. Γιατί εάν απελευθερώσουμε αυτά τα κεφάλαια σε αυτό το κλίμα στι αγορές, θα ενισχυθεί δυστυχώ η κατάσταση. Τώρα, αναφορές σε εποπτικές αρχές. Ε, το σκεπτικό εδώ πέρα είναι πως θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να περιοριστεί το βάρος της μικρές εταιρείε. Συμφωνούμε, αλλά βεβαίω υπάρχει και το τεστ του επίπεδου σημαντικότητα. δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα με το οποίο θα επιτρέψουμε στις μικρομεσαίες εταιρείες, εάν μπορέσουμε να τις ορίσουμε κατόπιν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, να αποφασίζουν για μια κάποια περίοδο να μην δίνουν κάποιες πληροφορίες σε εποπτικές αρχές. Στο πλαίσιο και εδώ πέρα της ε, φερεγγιότητας 2, όπου δίνουμε πολύ περισσότερο ρόλο στην αναφορά στις αρχές. Γι' αυτό θα πρέπει οι οπουδικέ αρχέ να έχουν τη δυνατότητα να ζητάνε πληροφορίε και αν δεν το κάνουν θα εξαναγκαστούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που θα απευθυνθεί στην ΕΟΠΑ και στα μέλη τη για τι πληροφορίε αυτέ. Οπότε αντί οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να εξαιρεθούν από κάποια πράγματα μπορούμε να εστιάσουμε στην σημαντικότητα για να μην αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια αιτήματα για πληροφορίε κατά το οποίο του κοστίζει. Και, να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, η Κομισιόν είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει, εσάς και τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής σας για να βρεθεί μια συμβαστική λύση για να καταλήξουμε σε αυτό για το οποίο και εσείς έχετε εργαστεί τόσο σκληρά και ο κύριος Μπάλτς επίσης και χαίρομαι για το ότι στηρίζουμε ακόμα την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπάλτς, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους του προλαλήσαντε αγορητέ για τις παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις που έκαναν. Και θέλω, αν γίνεται, κάποια θέματα να αναφέρω συγκεκριμένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω αναφέρθηκε, για το κείμενο για τι εκτελεστικέ διατάξει, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα μας τα υποβάλει τα σχετικά. Επανειλημμένα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή σήμερα θίξαμε αυτό το θέμα και ο Πίτερ Σκίνερ και η Πρόεδρος εξίσου και εγώ στι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις το έκανα. Το θεωρώ επιτακτική ανάγκη για την τελική φάση της έγκρισης Ψήφισή και Έγκριση, να γνωρίζουμε αυτέ τι εκτελεστικέ διατάξει από πλευρά κειμένου τη Επιτροπή. και χαίρομαι ότι τι επόμενε, θα έλεγα εν συντομία τρει εβδομάδε θα έχουμε την δυνατότητα αυτή. Τώρα, τι θα σημαίνει αυτό για εμά ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή από πλευρά χρονοδιαγράμματο. Θα πρέπει να δούμε σε εν χρόνο το τι θα κάνουμε. Είμαι ευγνώμων όμω για αυτή την ανακοίνωσή σα την κοινοποίησή σας. Δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να το τοποθετηθώ είναι το θέμα του Sunrise Clause που ως ρήτρα αναφέρθηκε από διάφορους προλαλήσαντες. Είμαι πολύ ανοιχτός για τη ρύθμιση αυτού του θέματος και σωστό, σωστά αναφέρθηκε ότι εδώ εμείς έχουμε μπροστά μας μια συγκεκριμένη δυναμική των πραγμάτων που εξελίσσεται. Και καλό αυτό. Και νομίζω, πιστεύω ότι θα βρούμε λύση για αυτό το ζήτημα. Τρίτο σημείο, από τη Σιλβί Γκουλά αναφέρθηκε. Επενδύσεις ε, σε μετοχές. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σπουδαιότατο θέμα. Πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ε, προανέφερε ότι εδώ θα πρέπει μια συνετή μεταβατική ρύθμιση να εξευρεθεί. Και εγώ συζητή σίγουρα με ιδιαίτερο τρόπο και σε, ε, με έκτακτο, σε έκτακτα μέτρα θα, μπορέσω, θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Τρίτο σημείο, το θέμα των ξεχωριστών συμφερόντων. Πράγματι, τι συμβαίνει εδώ. Μπορούμε να δούμε από κάποιες εξελίξεις και τοποθετήσεις με τροπολογίες που έχουν κατατεθεί αυτή την πτυχή. Είχα προναγγέλει εισαγωγικά ότι σκοπεύω να προσπαθήσω να εξεύρω συνετούς λογικούς συμβιβασμούς για τα διάφορα σημεία και γι' αυτό θα σταθμίσω και θα εξετάσω τα ξεχωριστά αιτήματα ή συμφέροντα με ξεχωριστό τρόπο. Και με τους σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να έρθω σε επαφή και να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Επόμενο σημείο, πέμπτο, για την ΑΙΟΠΑ. Πιστεύω ότι για μένα ως εισηγητή, αλλά και εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, είναι σαφές ότι ισχυρό ρόλο της ΑΙΟΠΑ επιθυμούμε να έχουμε όπως θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Και από πλευράς εξελίξεων βλέπουμε ότι υπέρ των ισχυρών εποπτικών αρχών και πρόπεση και πέρσι είχαμε τοποθετηθεί. Και εξού μετά από όλα αυτά πρέπει αυτή την έκθεση έτσι να την αντιμετωπίσουμε και να την δούμε. Να έχουμε έναν το δυνατόν ισχυρότερο, πιο ενδυναμωμένο ρόλο της ΑΕΟΠΑ. Έρχομαι τώρα στο θέμα των ε, προσεγγίσεων για τη σύνταξη εκθέσεων θέμα που έθιξε η Ελίζα Φερέιρα. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή τούτο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε πραγματικά πολύ προσεκτικά να διαφοροποιήσουμε ποιο θα υποβάλει ποιε εκθέσει, σε ποια πλαίσια και πώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μικρότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν και αυτές στην Ευρώπη θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα για αυτό το θέμα της προσέγγισης εκθέσεων και θα επιβαρυνθούν με αυτόν τον τρόπο υπέρμετρα. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και προσεκτικός να μην γίνει κάτι τέτοιο. Είχα και συχνές επαφές και συζητήσεις και μου είπαν οι μικρές ασφαλιστικές εταιρείες ότι αυτό είναι κέριο, κεντρικό θέμα και έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Ε, έβδομο σημείο που θέλω να αναφέρω δηλαδή τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ διαφωνώ ρητά. <clears throat> Δεν είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες τράπεζες και ούτε οι τράπεζες ασφαλιστικές εταιρείες αντίστροφα. Και γι' αυτό πρέπει πολύ προσεκτικά να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε, να δούμε πώς ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τομέα των ασφαλίσεων θα δημιουργηθεί, για τον ασφαλιστικό τομέα. Δεν πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση όπως την είχαμε στη ρύθμιση των τραπεζών. Μπορούμε να μάθουμε από αυτό το τομέα. Σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει. Αλλά να υπάρξει διπλοεπικάλυψη ή μίμηση και ε, με τον ίδιο τρόπο αντιγραφή αυτών που έγιναν στον τραπεζικό τομέα για τον ασφαλιστικό τομέα δεν συμφωνώ. Έχω προβλήματα με αυτό. Όγδο σημείο. Όγδο η τελευταία ε, παρατήρηση ρυθμίσεις με τρίτες χώρες. Εδώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τόνισε για άλλη μια φορά να έχουμε νόμιμα σωστά αιτήματα που θα διατυπώνονται προς τρίτες χώρες. Και όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο και από πλευράς εισηγητών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, σημαντικό σημείο. Το μάθαμε αυτό και το είδαμε στην οδηγία για τα FM. Είδαμε και Jean-Paul Gauzès πόσο δύσκολο ήταν να βρούμε μια σωστή διατύπωση. Και γι' αυτό είμαι και εδώ ρητά πάλι ανοιχτός και πρόθυμος για συζητήσεις και συμφωνίες. Συνοψίζω εν κατακλείδη. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ένας καλός συμβιβασμός είναι εφικτό και βρισκόμαστε στη σωστή πορεία θα έλεγα να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα με κάθε σαφήνεια να το εκφράσω, αυτό που η Κορίν Βόρτμαν Κόλ στην παρεμβασή τη είπε πιο πριν. Το ότι δηλαδή και για τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο ιστερότερα είναι πιστεύω σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει ένα σωστό συμβιβασμό που θα υιοθετήσει, ώστε με το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία να εγκριθεί και από την Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η επιθυμία μου ω ε, εισηγητή τι σε αυτή την επιθυμία έχω. Θέλω με τους χειώδεις εισηγητές και με τους άλλους να κατευθυνθούμε προς αυτή την πορεία. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα σημαίσιας διάταξης. Ε, μια ψηφοφορία η οποία όμως ε, περίτρα ρυθμίστηκε θα ξεκινούσε στις ε, ε, παρατέταρτο και βλέπω ότι δεν έχουν έρθει πάρα πολύ, άρα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να υπάρχει πληρότητα για ολομέλεια εδώ πέρα. Άρα έχουμε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή μας και μετά προχωράμε όλα σας στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ.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 Just. Have we got anything after votes, or then that's it? That's it. Two votes. Okay, okay, the sooner we start, the... Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε κιόλα. Οπότε, μπορεί κάποιο να πατήσει το κουμπάκι για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Right, test vote, please. Right. Right, press, press your yes button if you're... Πατήστε το ναι, εάν είστε χαρούμενοι. 33 βουλευτές έχουν ε, τις ε, κάρτες τους. Εάν κάποιος δεν έχει την κάρτα του, καλό να μα το πει τώρα. 36, 37, 38. you want try another seat? Okay. We've got, we've got some machines that aren't working. Κάποια μηχανήματα δεν δουλεύουν. Εδώ δηλαδή των αντιπρόεδρων. Και υπάρχει ένας παραπάνω από τους φιλελεύθερους. Α, δεν θα ψηφίσω εγώ λοιπόν. Βγάζω την κάρτα μου. It's easier if I don't have to vote. We've got 40 cards. 40. Συναδελφοί έχουν τις κάρτες τους, 33 μόνο έχουν ε, ψηφίσει. Μπορείτε να πατήσετε, σας παρακαλώ, το κουμπάκι. Doesn't work. Okay. Can you try, choose another seat? Καθίστε κάπου αλλού αν δεν δουλεύει. 38. Right, that's only Edward. Look. 38. Okay, so we've Και ο Εντουάρντ από τους σοσιαλιστές. Όλα εντάξει. Ωραία. Φαίνεται πως όλοι ήταν ικανοποιημένοι, αν και είχαμε και δύο εποχές. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση Ραμόν Τρεμόζα για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2010. Συμβαστική Α υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Β α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική C σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τα χέρια σας στο μέρος δεύτερο ξανά υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία του Sven Kigold την έχετε όλοι υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική δέλτα. Κάτι μου έχουν υπογραμμίσει εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εκτί, 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές καλύτερα να υπαλληθεύσουμε το δεύτερο μέρος της ε αρχίσει η ψηφοφορία. Δουλεύουν λοιπόν τα πάντα πέρα στις ε, ψηφοφορίες δεχτεί. 23 υπέρ, 16 κατά, 70 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, σήμερα μου το βλέπω να επαληθεύσουμε την 70. Ψήφισαν όλοι. Τέρας. Δεκτή. 22 έναντι 20. 71 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Ορίστε. Ε, εμένα έτσι μου φάνηκε. 72. Λοιπόν. Υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έγινε δεκτή να επαληθεύσουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Καταπίπτει. Με ισοψηφία. 73 υπέρ. Κατά. αποχές. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 τροπολογία. Α, μια στιγμή. F α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην συμβαστική G, μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος. όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 91 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Μέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε Τροπολογία 92 υπέρ. Ενενήντα δύο υπέρ, κατά. Δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια, να επαναλάβουμε την ψηφοφορία και πάλι. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε τώρα, εντάξει. Η 91 κατέπεσε, εντάξει, με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 94 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε, ψηφίζουμε την 94, άρχεται. Yeah, I think it's carried because of... Νομίζω είχε εγκριθεί Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε όμως, μάλιστα. Τροπολογία 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή εγκρίθηκε. Συμβιβασμός GA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός H υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός I υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός J υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός K υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 129 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. 130 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. Παράγραφος 14. Προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός L. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές 143 έως 147 ομού όχι ε όσοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 145 υπέρ κατά αποχές όχι, προσέξτε, δεν γίνεται. Ρώτησα να ψηφίσουμε όλες, είπαν όχι. 145 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. 146, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εν α υπέρ, εν ε υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε, θα αναβάλουμε τώρα σε σχέση με την 155 και τα λοιπά. Φτάνουμε στον συμβιβασμό Κιούνα. το ξέρετε, δεν το έχω ξεχάσει. 156 τώρα υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Ο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και αυτό. Συμβιβασμός, όχι, τροπολογία 169 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 169, έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη ισοψηφία 21-21. 170 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός πι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός PA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε 184 υπέρ α, συγγνώμη, ε, κατέπεσε αυτή μάλιστα πάμε στην 185 185 υπέρ κατά να, επαναλάβουμε πάλι 185 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός Q σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα παρακαλώ του συμβιβασμού Q. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και τώρα η 155 καταπίπτει γιατί συμπεριλήφθηκε στο συμβασμό Q και καλύφθηκε έτσι. Συμβασμός 190 τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Α σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα του συμβιβασμού R άρχεται. Πρώτο τμήμα συμβιβασμού Α άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πρώτο τμήμα του Α. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. Ισοψηφία καταψηφίστηκε 21-21. Να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα τώρα. Καταπίπτει λέγεται στην πρόεδρο. Καταπίπτει. Γιατί. Δεν βλέπω γιατί. Λοιπόν. Εισηγητά. Νομίζω το δεύτερο τμήμα μπορεί να ψηφιστεί, να τεθεί σε ψηφοφορία. Ακόμα και αν καταψηφίστηκε το πρώτο. Έτσι, λοιπόν, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 204 τροπολογία υπέρ. Α, κατέπεσε αυτή εντάξει κατέπεσε, πάει αυτή. 206 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται, ψηφίζουμε την 206. Ελέγχουμε την 206 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Καταψηφίστηκε. Η 207 υπέρ. Κατά. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 207. 207 ηλεκτρονικά. Δεν βλέπω και δεν είναι ευδιάκριτο το αποτέλεσμα με τα χέρια που σηκώσατε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρι... Απορρίφθηκε, διορθώνει Πρόεδρο. Απορρίφθηκε. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι, λυπάμαι, πρέπει να ελέγξουμε την 208 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα που πρέπει να ψηφίσουν. Πατήστε το κουμπί σας τώρα, θα λήξει η ψηφοφορία. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, έληξε, απορρίφθηκε λοιπόν. Τροπολογία 209, υπέρ. Κάτα. Αποχές, απορρίφθηκε. Ποιαν είπα? για τη 205 Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η 205 λοιπόν. Ως είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός S. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 216 υπέρ Α, κατέπεσε. Ωραία. Λυπάμαι. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι στο γκρι χρώμα. Φαία τροπολογία. 217 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. Άρα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 217 και άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι καταψηφίστηκε. Ισοψηφία 21-21 καταψηφίστηκε. 218 υπέρ. Κατά αποχές. Πώς ψήφισαν οι σοσιαλιστές για την 218 υπέρ, υπέρ, εντάξει ευχαριστώ, εγκρίθηκε λοιπόν. 219 κατέπεσε, 220 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Διαμαρτυρίες. Να ελέγξουμε την 220. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία 220. ...220 λοιπόν ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα καταψηφίστηκε με μία ψηφοδιαφορά μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είχα δίκιο εσείς άδικο. Λοιπόν, τέλεια. Τροπολογία, τροπολογία 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ωραία. Λοιπόν, αιτιολογικές. Στα εκτιμώντας, στα εκτιμώντας, ομού να τα πάρουμε. Έχω συν και πλήν όμως τον πίνακα παντού, δεν γίνεται όλες από κοινού. Λοιπόν, η 1 και 2 εκτιμώντας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Εκτιμώντας τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εκτιμώντας τέσσερα μέχρι το επτά ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. Πάμε στον συμβιβασμό τι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβιβασμό U υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στον συμβασμό W υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε θα ψηφίσουμε τώρα στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε συνολικά ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 35 υπέρ, 4 εναντίον, 3 αποχές. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή.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 Okay, is everybody ready? This is the vote on. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, ψηφίζουμε το σχέδιο γνωματοδότηση του Αλφρέντο Παλώνε για τη νέα στρατηγική πολιτική καταναλωτών. Λοιπόν, να κλείσει η προηγούμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, έχω κατάλληλε ψηφοφορίε. Yeah, I... Yeah, Right. Λοιπόν, τροπολογία 1, ε, ναι, προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Καταρχάς λοιπόν να ακούσουμε την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, σε δύο μέρη. Το πρώτο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, ε. Λοιπόν, επανέρχομαι αφού πέρασε η προφορική τροπολογία, ξεχνάμε τα επόμενα. Παράγραφος 2. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σύγχυση. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν αρκεί ανάταση χειρών. Λοιπόν, εγκρίνεται. Άρα δεν έχουμε ξεχωριστή πληροφορία συνέχεια, αφού εγκρίθηκε αυτή. Παράγραφος 3. Στο κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 όπου και αν έχει πάει και που βρίσκεται. Λοιπόν, τροπολογία 7 σε δύο τμήματα. Το πρώτο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική C, σε άλλη σελίδα, υπέρ, κατά, μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή υπήρχε μια προφορική τροπολογία του εισηγητή που ξεχάσαμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Προφορική από Όχι, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτή την τροπολογία. Είμαι αντίθετος σε αυτή την τροπολογία, γιατί πιστεύω ότι είναι συμπροματική με την συμβιβαστική 8 δέλτα. Για μένα λοιπόν είναι σαφές ότι είναι αντίθετο στην προηγούμενη προφορική τροπολογία. Καλώ. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν αυτή την προφορική τροπολογία του εισηγητή, άρα ψηφίζουμε το κείμενο σε τρία τμήματα. Το πρώτο, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Το τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πηγαίνω στην συμβιβαστική σηματάφα αντιπρό F, σελίδα 11, σε δύο τμήματα. Πρώτο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι επίσης εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική G Σελίδα 13. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική age στην ίδια σελίδα, σε δύο τμήματα. Το πρώτο, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, επίσης εγκρίνεται. Και τώρα, είμαστε τελευταία στο σύνολο του κειμένου, κατόπιν των όλων τροποποιήσεων, ηλεκτρονική ψηφοφορία. στις ψηφοφορίες. 38 υπέρ και 2 κατά καμία αποχή. 36 μάλλον υπέρ επί 38 ψηφισάντων. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ολοκληρώνουμε τη συνεδρία αυτή, τη συνεδρία Ιεγκέρος. Ευχαριστώ τους πάντες.